It's a problem of those who are not here. Good morning, everybody. We have very few time. We have one. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι επειδή έχουμε πολύ δουλειά μπορούμε να αρχίσουμε. Τι να σα πω, schön, καιρός, καλή σα μέρα. Για να ξέρετε αν είναι ένα μέρο το ακουστικό δηλαδή, έχει τίποτα άλλο. Ναι, είναι, είναι. Λοιπόν, χθε το βράδυ είχαμε μια συνεδρία των συντονιστών. Τα αποτελέσματα τα έχετε λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρακαλώ να ασχοληθείτε με αυτό και να μας πείτε αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε. Ωραία. Περνάμε στην μαρμοδότηση της Ρόζα Κόμισα του Τόντσαν. Α, όχι, κυρία Παλιαδέλη, συγγνώμη. Της κυρίας Παλιαδέλη την έκθεση έχουμε αρχικά. Συγγνώμη. Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτού, κυρία Παλιαδέλη. Παρακαλώ. Short, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που μου δίνει την ευκαιρία να εργαστώ για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τονίσω πόσο καλή συνεργασία είχαμε με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές και τους συναδέλφους μου και το Συμβουλίο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, μετά από αυτές τις ευχαριστίες μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. Έχετε τις κάρτες σας, τις ε, κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας. Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. της 10 κατά, συγγνώμη, 15 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. Das ist komisches Ding Just a moment, I have to look here. Μια στιγμή να δω τι γίνεται εδώ, λέει η πρόεδρος. Μάλιστα. 5 υπέρ, 10 κατά. Απορρίπτεται. Εσύ τι ήσουν υπέρ κατά. Υπέρ. 6 υπέρ 10 κατά. So once again that Mrs. Palliate... Η κυρία Παραδέλη πάλι 6 υπέρ 10 κατά λοιπόν στην έκθεση αυτή επί των Μα écoutez, êtes là, attends, vous avez du Ακούστε, σας έδωσα χρόνο να ψηφίσετε. Λοιπόν, 7 υπέρ 11 κατά. Τελειώνουμε. Εδώ κλείνουμε. Άστρο 2. Τροπολογία 60. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 61. Αποσύρθη. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 απεσύρθη 64 απεσύρθη 7 υπέρ κατά να ελέγξουμε άρχη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 12 προς 12 απορρίπτεται 65 απεσύρθη 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 καταπίπτει. 66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε. Άρχισε ψηφοφορία. Σκεσλώσεν. Πέρας. 12 προς 13. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Για να ελέγξουμε, για την 70 ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. 15 υπέρ 12 κατά. Συγγνώμη, εγκρίνεται πράγματι. Εβδομήντα ένα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, δέκα, υπέρ, κατά, αποχές, α, εγκρίνεται, έντεκα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 78 Άχι ψηφοφορία Geschlossen. Πέρας. 16 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17. Α, καταπίπτει. Α, 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. 15 προς 10 εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχη ψηφοφορία. πέρες ψηφοφορίας. 81 εγκρίνεται. 14 προς 13. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Για την 85. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 15 προς 12. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, καταπίπτει. Α. 89. Ναι, 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν, δεν, δεν είσαι στη σωστή θέση, γι' αυτό με μπερδεύετε. Ένα από τους αδέλφους του ΕΛ κάθεται αριστερά και μπερδεύομαι. Ο νέος συνάδελφος από την Ουγγαρία. Καλωσορίσατε, ορίσατε. Αλλά εδώ καθόμαστε σωστά. Δεν βρεις θέση ε. Κάτσε κάπου τέλος πάντων. πίστ. Irgendwo dahin, ja. Nimm das von Βερονίκ, μπορείς παρακαλώ να βοηθήσεις τον κύριο. Ωραία. Μπράβο. 90 υπέρ. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 και 92 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος. Άχι ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρασε ψηφορίας 17 προς 11 εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. 26 προς 1 εγκρίνεται. Γιατί δεν σηκώσετε τα χέρια σας. Υπάρχει μια καθυστέρηση συνήθω από την ώρα που το λέω μέχρι τι και Τέλο πάντων, 99 υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 100 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά έλεγχος για την 102 πέρας 14 προς 13 εγκρίνεται 104 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά, πέρας, εγκρίνεται. 16 προς 11, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχισε ψηφοφορία για την 105. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 προς 8. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Ενεκρίθη 15 προς 13. Ένας πράσινος βουλευτής είναι παραπάνω από που χρειάζεται. Να είσαστε υπέρα μα θέλετε, να μην ψηφίζετε. Green. Ποιοι είναι οι πράσινοι εδώ. Γιουνκέρας και πριν από Η κυρία Τρούπερ, ας μην ψηφίζει. Κατ' εξαίρεση βέβαια. Was Δεν είχαμε τίποτα με διαφορά μια ψήφου. Στην αρχή αρχή ίσως. Που είχαμε μία υψοψηφία. Could you use your micro? Παρακαλώ μικρόφωνο. Δεν ακούγει αλλιώ. Εκτός μικρόφωνο. Είσαστε σίγουροι ότι η διαφορά δεν ήταν... Σε αυτό εδώ το τελευταίο να το ελέγξουμε. Ποιο θέλετε. 106. Ωραία. 106. Ποιος είναι υπέρ της 106. Κατά. Ναι, ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 προς 13. 12 προς 13 απορρίπτεται. Δεν λειτουργήσε. Και 13 προς 13 απορρίπτεται. Παρακαλώ. Er δεν έχει κάρτα και είναι υπέρ. Άρα 14 προς 13 είναι κρίθη. Nein, bitte. Ο νέος συνάδελφος από την Ουγγαρία δεν έχει κάρτα. Καταλάβατε. Και πρέπει να το μετρήσω. Και ο Κάμερτας η κάρτα του δεν λειτουργήσε. Θα πρέπει να τον υπολογίσουμε επίσης. Και φτάνουμε στο 12 υπέρ 14 ε, υπέρ και 13 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Ωραία. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πού είχαμε μείνει. Στο 108. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχη ψηφοφορία. It's closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Καλά, καλά. 110 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία σου. Ναι, εγκρίνεται. 18 προς 11. Προφορική τροπολογία της κυρίας Ράνερ. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. 11 προς 13 απορρίπτεται. 111. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Α, τι. Καταπίπτει. Α, καλά. Καταπίπτει. Ωραία. 27 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. η Φορεία Πέρας. Απερίφθη. 13 προς 14. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 36 ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας πληροφορίας. απορρίπτεται λέει πρόεδρος α όχι όχι εγκρίνεται 16 υπέρ 12 κατά πρέπει να σας έχω και εσάς εκεί υπόψη μου Ωραία. 126 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 15 προς 12 37 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 37 πέρας 15 προς 11 εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ποιο να ελέγξουμε. Τη 42 ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρασε. <laughs> 29 υπέρ, 0 κατά. Μα υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση. Yeah. Should I say it in English? Ja, ich hab's verstanden, ja. Ich mach's doch nur euch zu. Εγώ βιάζομαι γιατί και εσάς. 43. Υπέρ, κατά. Λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 31. 131 μάλλον, υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει. Α, να μου το πείτε αμέσως παρακαλώ. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 54 της ψηφοφορίας 19 προς 9 εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά να ελέγξουμε εντάξει 4 ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας Εγκρίνεται 28 προς 2. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στο τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 28 προς 0. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Παταδέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Καμερέβερτ. Θέλει το λόγο, κυρία Καμερέβερτ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κατά βάση να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνεργάστηκαν. Εδώ ήταν πολύ σκληρό το έργο. αλλά άμα το εγκρίνουμε νομίζω ότι θα έχουμε ε, βελτιώσει την πρόταση οδηγία που μα έχει υπευλήθει. Θα ήθελα ευχαριστήσω ιδιαίτερα σκιώδη σκιώδες του ε, συντονιστέ και τον Στέφανη, την Στεφανή Πιεζόλη που είχε πάρα πολύ δουλειά τι τελευταίε μέρε με τη λίστα τη ψηφοφορία. Ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Τίτλ. Amendment 80. Wer ist dafür? Το 80, υπέρ. Κατά. Ξανά. Ποιο είναι υπέρ τη 80. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 12. Α, 13 υπέρ. Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, 12 λέει διαγραφή, διαγραφή. Ναι, συγγνώμη. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ Εάν το εγκρίνεται θα διαγραφεί αυτό. Ε. Α? 17 έχουμε λοιπόν. 17 έχουμε τώρα. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Γιατί 17. Πέρας. 16 προς 13 εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122. Υπέρ. Κατά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 αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ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

Η Οζέπλε παρεμβάσει εκτό μικροφώνου, δυστυχώ. So, mein Gott, nochmal. Also 141. So, once again, because you were... Λοιπόν, 141 ξανά γιατί έκανε λάθος. Δεν ξέρω προς τα ποιο κατεύθυνση έκανε λάθος, πάντως λάθος. 141. Ωραία. Πέρας. 12 προς 16. Και μεσάς 17. Απερίφθη λοιπόν. 12 προς 17. Α, έχεις κάρτα. Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Απορρίπτεται πάντως. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωτο. 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προβολική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχή. Προβολική τροπολογία, υλικό καλπέλες. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 προς 16. 56 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχισε ψηφοφορία. Για την 56 πέρας. Εγκρίνεται. 25 προς 6. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 57 παρακαλώ Πέραση ψηφοφορίας Δεκαπέντε προς 16 απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές μάλλον η ήθελα για να ελέγξουμε για την 156 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα έχουμε ένα σοσιαλιστή που περισσεύει. One socialist has to check. Mr. you forget to... Και με ψηφίσετε. Παρακαλώ μη φύγετε όμως, θα σας χρειαστούμε. 58 υπέρ. Κατά. 58 λέω υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Das kann ja nicht wahr sein. 58. 58. 58 είπα. The wall is closed. The which is the, the number? 158. Ja, Moment. Okay, okay. Das Sekretariat hat mir... Okay. 158. Δεν φταίω εγώ πάντα, η γραμματεία δεν μου τα σωστά 158. 158. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. 14 15. Απορρίπτεται λοιπόν. 159 υπέρ κατά αποχές άρχιτε ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 από 14 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 η τρίτη παράγραφος έχει αποσυρθεί. Ωραία. Η κυρία Μακλάκιν θέλει να αποσύρει την τρίτη παράγραφο, αλλά το υπόλοιπο της τροπολογίας παραμένει. Λοιπόν, πώς είναι υπέρ, λέει η πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχιτε ψηφοφορία πέρας 14 προς 15 απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 It was not adopted, it was rejected. Απεσύρθη 61 λέει η πρόεδρος. Η παρέμβαση δυστυχώ ήταν εκτός μικροφώνου. 166 είμαστε τώρα, υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές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 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές Έχω κάποια προβλήματα με τους φιλέτερους, να τα πάμε από κοινού δηλαδή. Λοιπόν, 67 έως 76, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 176 λοιπόν <clears throat> υπέρ κατά να ελέγξουμε την 176 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 14 προς 15 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν 178. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτο. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απαραίτητε. 12 προς 18. Συμβαστική 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 και 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 102 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Για την 102 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 15 προς 14. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. 25 προς 0. Ευχαριστώ. Δύσκολα πολύ καλά. Συγχαρητήρια κυρία Καμερέβερτ. Και ευχαριστούμε και τους Κιώδης. Τελειώσουμε πριν από τις 10. Ρόζα Φοντούνουν Χοενστάιν. Θες να σου δώσω το λόγο, Ρόζα. So, um... Thank you very much for the... Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Αυτό το έγγραφο σε αυτή την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτικών, όπως επανειλημμένα είπαμε, δημιουργεί πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα και όχι μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περιμένουν αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει κάτι να προκύψει πολύ πιο φιλικό στον πολίτη από ότι το έγγραφο της Κομισιόν και αυτό το έγγραφο προτείνει μια στάση πιο ανοιχτή και απλουστεύσαμε τις άλλες διαδικασίες και υπάρχει η ψήφιση του σημείου 59. Εδώ ζητήθηκε μια συνάδελφο να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Έγγραφο όχι για εμάς, αλλά για τους πολίτες και γι' αυτό παρακαλώ να επιψηφίσετε και τα δύο τμήματα του 59. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ Ρόζα. Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό λύση, γητρία. Μισό, μισό λεπτό. Α. Πέρασε ψηφοφορία. 7 προς 22 με τη Ρόζα, γιατί δεν πρόλαβε η Ρόζα να ψηφίσει. Ωραία. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Ακαταπίπτει. Α, ναι, ναι. Στο 61 περνάμε. Πολύ ωραία. 61 λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ Α, εδώ έχουμε τα δύο τμήματα Πρώτο τμήμα υπέρ vote both. Wir stimmen beide. No, it's okay. We have to vote. Ναι, ναι, πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, 59 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Όχι. Αχ, όχι. Στην έξι πάμε. Συγγνώμη. Έξι λοιπόν. Έξι. Υπέρ. Κατά. Απαχές. Εγκρίνεται. Εξταπέντε. πέντε. Απεσύρθη. Εξτεφτά. εφτά. Υπέρ. Εξτεφτά. εφτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 και 68 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. He missed his traffic this morning. He had to walk, and now he is really tired. So, okay. I'm. Έχασε το λεωφορείο, το πρίξε με τα πόδια, φαίνεται και είναι πολύ κουρασμένος. Ποιος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 έχει αποσυρθεί 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά για να ελέγξουμε για την 72 πέρα ψηφοφορίες απορρίπτεται 9 προς 20 74 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται 75 α όχι καταπίπτει 9 9 9 9 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται δώδεκα δώδεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ογδόντα, ογδόντα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ, κατά ξανά 81 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 81 ηλεκτρονικός έλεγχος <coughs> πέρας 16 προς 14 εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. 86 γνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 ταυτόσημη. 84 και 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 καταπίπτει. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά έχει καταπέσει α ναι ναι 16 λοιπόν κατέψει 92 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 16 πέρας 20 προς 10 εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά είναι νομίζω να ελέγξουμε την 106 Πέρας. 20 προς 8 είναι κρίση. 18 υπέρ. Κατά. Ξανά. Ποιος είναι υπέρ της 18 παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 31 και 33 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 38 ελέγχουμε πέρας ψηφοφορίας 20 προς 9. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 46 η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 21 προς 8 47 υπέρ κατά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 Το δικό σας δεν Α, 29 λοιπόν υπέρ. 30, 30. 30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω ότι αυτό το νέο μέσο θα μπορέσει να είναι πολύ χρήσιμο. Έχω αμφιβολίες εγώ προσωπικά, αλλά θα δούμε. Ολοκληρώσαμε τώρα τις ψηφοφορίες. Σε τρία λεπτά θα αρχίσουμε την ακρόαση. Παρακαλώ όλους τους αδέλφους να παραμένουν εδώ σε, στην αίθουσα. Έχουμε πολύ διακεκριμένους προσκεκλημένους για την ακρόαση. Και δεν θέλω να μην είσαστε παρόντες. So for everyone who is interested, there is a 1G3. So if you don't... Εάν δεν βρείτε θέση να κάτσετε εδώ, να πάτε στο 1G3 όπου μπορείτε να ακούσετε. Καλημέρα στους προσκεκλημένους μας. Ολοκληρώσαμε την ψηφορία because... που ήταν πάρα πολύ δύσκολα να τα καταφέρουμε γιατί υπήρχαν επίμαχα σημεία και θα σας τα πω στα αγγλικά γιατί προετοιμάστηκα να τα πω στα αγγλικά και συμπαθάτε μέσα νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα μας γιατί συνήθως το κάνω. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το πόσο αξίζει ο πολιτισμός σε σχέση με την ε, πολιτική μας ευρωπαϊκή ταυτότητα και σε σχέση με τον κινηματογράφο. Αυτό όλοι μπορούν να το διαπιστώσουν. Αν πάτε στον τρίτο όροφο θα δείτε ε, ότι είναι τιμόμενος αυτές τις μέρες ο κινηματογράφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε αυτά τα ε, βραβευμένα έργα τις επόμενες εβδομάδες τα οποία εκεί παίζονται και προσέξτε και στο θα ψηφίσετε για αυτά τα έργα όμως όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια αυτού του βραβείου Lux σε σχέση με το κινηματογράφο οπότε και για αυτό το λόγο καλέσαμε αυτούς ε, τους εξαιρετικούς μας φιλοξενουμένους, αλλά πριν τους το λόγο επενθυμίζω σε όλους ότι εδώ και πάνω από 10 χρόνια δίνουμε μάχη για τον κινηματογράφο με το Media Procam. 8 χρόνια δηλαδή, που σημαίνει Media Program σημαίνει προώθηση και διανομή ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων. Και θυμάμαι ότι ακόμα και στο τέλος του προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας ε, που κάναμε ε, πάρα πολλά βήματα πρόοδου με τον συνάδελφο Γερόνιμη και είχαμε μετά το Media Mundus 2011-2013 θα πάει αυτό το πρόγραμμα κάτι το οποίο θα τρέξει σε όλη την Ευρώπη. Επίσης μιλούμε για την ψηφιοποίηση και χθες ήρθε η Επίτροπος η κυρία Βασιλείου η οποία είπε σχέθη ότι θα βοηθήσει για την ψηφιοποίηση και των κινηματογραφικών έργων όσον αφορά κάποιους ε, πόρους και όσον αφορά την ε, αυτές τις ε, ε, εκπομπές μέσω του δικτύου EBD. Ο κύριος Βέντες κάθεται δίπλα μου με μεγάλη μου χαρά. Τι να σας πω για αυτόν, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Είναι ένα σκηνοθέτης διάσημος, αλλά επίσης είναι και ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. και παρίσταται και τον συνοδεύει και ο γραμματέας της Ακαδημίας αυτής. Και έχουμε αυτά τα ευρωπαϊκά Όσκαρ, τα οποία πανέμονται κάθε χρόνο. Πέρσι αυτό έγινε στην Πολιτική της Ευρώπης, στο Έσεν, κοντά στο Μπόχουμ. Στο Μπόχουμ, είναι στην περιοχή του Έσεν. Και έχουμε και κάποια άλλα επιτεύγματα όπως αυτή την ε, ομάδα προβληματισμού για την εικόνα της Ευρώπης, την εικόνα στην Ευρώπη. Επομένως, βοηθάει πάρα πολύ όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Είναι και φίλος του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προηγούμενου και του νυν Πρόεδρων του Κοινοβουλίου, του Πέτριν και του Μπούζεκ. Αυτά για τον πρώτο μας ομιλητή. Οι υπόλοιποι θα είναι σκητάλη στη συνέχεια, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και τώρα σας δίνω το λόγο κύριε Βέντερ. Καλημέρα σας. Σας απευθύνουμε πραγματικά ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που εκπροσωπεί 240 ε, επαγγελματίες ε, του χώρου του κινηματογράφου. Ε, τον Μάιο του 2009, 20 από αυτούς τους ε, ε δημιουργούς ε, δημιούργησαν ένα think tank υπό την ε, εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σκεφτούν και να προβληματιστούν όλοι μαζί για την εικόνα της Ευρώπης. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εντοπίσει η ομάδα αυτή τα κενά ή τα προβλήματα αυτής της εικόνας. Οι σημερινοί Ευρωπαίοι βλέπουν την Ευρώπη κυρίως ε, σαν μια πολιτική, τεχνική, γραφειοκρατική δομή που ενδιαφέρεται περισσότερο για τα οικονομικά θέματα. Η διοίκηση της Ευρώπης έχει γίνει η εικόνα της Ευρώπης. Ήταν ε, ένα απογοητευτικό συμπέρασμα αυτό και είναι η εξήγηση για τον τρέχοντα ευρωσκεπτικισμό θέματα εικόνας και ταυτότητας ε, συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Το να ξέρει κανείς ε, ποιος είναι σημαίνει να ξέρει σαν τι μοιάζει και αντιστρόφως. Το πώς βλέπεις καθορίζει το πώς γίνεσαι ορατός. Κάναμε μια πολύ ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ε, ε, Βαρόσο που ε, συζητάει μαζί μας σχετικά με το πώς αυτή η απογοητευτική εικόνα για την Ευρώπη μπορεί να βελτιωθεί και το συμπέρασμα προήλθε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μας στην συναισθηματική πλευρά της Ευρώπης. Ίσως δεν σας πάρει έψη να ακούσετε ότι οι 20 αυτοί κινηματογραφιστές του Think Tank ε, είδαν το δικό τους ε, μέσο, το φιλμ δηλαδή, το κινηματογράφο, σαν τη λύση για το πρόβλημα. Για να μην πω σαν ένα μυστικό όπλο για την επίτευξη αυτής της αποστολής. Θεωρούμε το κινηματογράφο σαν ένα από τα πιο κατάλληλα μέσα για να βελτιωθεί το συναισθηματικό έλλειμμα στην πρόσληψη της Ευρώπης. Ο πολιτισμός συνολικά και με την ευρύτερη έννοια είναι ακριβώς η κόλλα που δημιουργεί τις ταυτότητες και καθορίζει την ε, ε ψυχή της Ευρώπης. Και ο κινηματογράφος έχει προνομιούχα θέση ε, από αυτή την άποψη. Είναι ένας ε, δημοφιλής τρόπος για να διαδοθούν ε, κοινωνικά, ε, ηθικά και πολιτιστικά μηνύματα. Ε, δημιουργεί ταυτότητες σαν κανένα άλλο μέσο και προσδιορίζει συναισθηματικές και γνωστικές διασυνδέσεις. Δεν προβάλλει μόνο εικόνες το φιλμ, αλλά αντικατοπτρίζει την εικόνα της πραγματικότητας την ίδια και παρουσιάζει όλους τους τα, τα ήθη και τα έθιμα, τις ελπίδες, τους φόβους. Και πάνω από αυτό διαμορφώνει τις αξίες ο κινηματογράφος και επηρεάζει τάσεις, ελπίδες και φόβους. Οι, οι ταινίε πρακτικά επινόησαν το αμερικανικό όνειρο. Μπορούν να κάνουν θαύματα για την εικόνα τη Ευρώπη, αρκεί μόνο η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει περισσότερο, να αξιοποιήσει περισσότερο τον ίδιο τον κινηματογράφο της, για την εικόνα τη και για την αυτότητά τη. Αν δεν ήταν τόσο επιφυλακτική ε, η Ευρώπη, ε, τόσο ντροπαλή όσον αφορά τα μεγαλύτερα πολιτιστικά της προσόντα και ιδίως το κινηματογράφο της. Αν πάτε στα μεγάλα μουσεία, σε όλη την Ήπειρο, Κάθε πρωί θα συναντήσετε πάρα πολλά παιδιά που μαθαίνουν ε, με αυτόν τον πολύ ε, σημαντικό τρόπο για την τέχνη. Η τέχνη και η ιστορία της τέχνης είναι βεβαίως η, ε, είναι μέρος της, ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τα παιδιά το ξέρουν αυτό. Άμα πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο θα δείτε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία τα περισσότερα από αυτά ευρωπαϊκά. Λογοτεχνία, θέατρο, ε, ποίηση, όλα αυτά είναι αφιζήτητα μέρος της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. αν σε ένα βιβλιοπωλείο το 50 ή το 80% των βιβλίων ήταν αμερικάνικα, αυτό θα δημιουργούσε τεράστια κατακραυγή. Το ίδιο και Στι συναυλίε. Κοιτάξτε όμω τι γίνεται κινηματογραφικέ αίθουσε σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία κατακραυγή. Μερικές φορές οι μισέ οθόνες σε μια ολόκληρη χώρα ε, καταλαμβάνονται από μία και μόνο ταινία. Προσπαθήστε να το μεταφράσετε αυτό ε, στα, στο επίπεδο των μουσείων, των βιβλιοπολίων ή των αιθουσών ε, συναυλιών. Δεν θέλω να παραπονεθώ όμως, γιατί ε, πρέπει να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές ταινίε είναι σε πολύ καλή κατάσταση συνολικά, ε, χρησιμοποιούν ε, το συνέστημα, το χιούμορ, ε, την επινοητικότητα. Κοιτάξτε τις ταινίε. Πάντα να δείτε τις ταινίε που είναι υποψήφιες για το βραβείο Λουξ. Ε, οι ευρωπαϊκές ταινίε καταλαμβάνουν ή το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο, ανάλογα με τη χώρα, των ε, κινηματογραφικών αιθουσών σήμερα σε όλη την Ευρώπη, που 20 χρόνια πριν κάτι τέτοιο θα το θεωρούσαμε ε, α, αδύνατο να συμβεί. Α μην παραπονούμαστε λοιπόν. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και για το παρελθόν και για το παρόν του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Είμαι εδώ να μιλήσω όμως για το μέλλον, αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Θέλω να μιλήσω για τα παιδιά, τα μικρά παιδιά και τους εφήβους. Το μελλοντικό μας ακροατήριο βεβαίως. Αλλά πάνω απ' όλα ε, δεν είναι μόνο το μελλοντικό μας κοινό, αλλά είναι οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι. Για αυτό το μελλοντικό κοινό η επιλογή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου δεν υπάρχει πια. Για αυτούς κινηματογράφος ήσουν blockbusters. Μια γιγαντιαία παγκόσμια ε, βιομηχανία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και εστιάζει πάνω στα παιδιά με, μεγάλα, με, με ένα τεράστιο οπλοστάσιο. Γι' αυτό στα μάτια τους ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος σχεδόν δεν έχει καμία ελπίδα. Γίνεται ένα είδος που απειλείται από εξαφάνιση. Είναι γεγονός ότι ο κινηματογράφος μας συνολικά κατευθύνεται, ε, απευθύνεται μάλλον σε πιο ενήλικο κοινό. Είναι το slow food σε σχέση με το fast food και ξέρουμε ότι το slow food είναι το καλό φαγητό. Αλλά το γεγονός είναι παρόλα αυτά ότι χάνουμε το νεανικό κοινό. Δεν πρέπει όμως να είναι τα πράγματα έτσι, πιστεύουμε. Είναι πράγματι απαράδεκτο αυτό όταν ε, διαπιστώσει κανείς ότι η παρακμή για την οποία μιλάω είναι εκπαιδευτική, είναι παρακμή της παιδείας. Ένα κοινό, έστω και με ε, αμυδρή ε, γνώση της ιστορίας του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, θα έπρεπε και θα ήταν σε θέση να επιλέξει διαφορετικά, θα, έκανε, θα έπαιρνε διαφορετικές αποφάσεις το γούστο μπορεί να διδαχθεί. Όμως, η έβδομη τέχνη διαδραματίζει έναν ε, ελάχιστο ρόλο, αν όχι και μηδενικό ρόλο, στο σχολικό πρόγραμμα όλων των ε, σχολείων μας. Δεν αξιοποιούνται κατά κανέναν τρόπο οι εξαιρετικές ε, ε ιδιότητες που έχει ο κινηματογράφος σαν εργαλείο εκπαιδευτικό. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να διδαχθεί και να τη μάθει κανείς. Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τα οπτικοακουστικά μέσα. Τα παιδιά κάθε μέρα ε, αφιερώνουν σημαντικά περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση ή στο κομπιούτερ παρά πάνω σε ένα βιβλίο. Όμως η ε, οπτική γλώσσα ε, είναι μόνο κάτι το συμπληρωματικό και δευτερεύον στο σχολείο, αν υπάρχει καθόλου. Είμαι εδώ σήμερα ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου για να επιβεβαιώσω σε αυτούς που έχουν τα πολιτικά μέσα και την πολιτική εξουσία ε, για να δώσουν στην εικόνα του κινηματογράφου μεγαλύτερη σπουδαιότητα μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από ό,τι έχει μέχρι σήμερα. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από εικόνες ε, παντός είδους και έχουν ε, σημαντικές ε, δυνατότητες να μάθουν τη γραμματική και το λεξιλόγιο αυτής της γλώσσας. Πολλοί από εσά και εμείς σίγουρα έχουμε δίκιο να ανησυχούμε για το γεγονός ότι τα βιβλία χάνουν την έλξη τους απέναντι στα παιδιά. Δεν είναι όμως ε, ακόμα πιο απογοητευτικό αν, ε, δεν, αν, παρετηθούμε από την ε, επιθυμία μας να διδάξουμε την γλώσσα της εικόνας στα παιδιά ή αφήσουμε σε άλλους να το κάνουν αυτό. Η κινηματογραφική παιδεία, ο κινηματογραφικός αλφαβητισμός είναι κάτι που πρέπει να μπει στην ατζέντα των Υπουργών Πολιτισμού με σκοπό η τέχνη ε, και η λογοτεχνία του κινηματογράφου ε, να γίνει ένα ε, σταθερό κομμάτι του σχολικού προγράμματος και όχι μόνο να χρησιμοποιείται σαν κάτι το δευτερεύον. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι ένα όραμα δεν είναι το ίδιο με την πολιτική πραγματικότητα. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά των ίδιων των κρατών μελών σαν ανταπόκριση ε, στην πρόκλησή μας, πολλοί υπουργοί σε όλη την Ευρώπη ε, είναι πρόθυμοι να μας, ε, και μας γνωστοποιούν ότι εκτιμούν όλους ιδιαίτερος την έκκληση μας αυτή και ότι έχουμε απολύτως δίκαιο σε αυτά που λέμε. Και κατέστησαν σαφές ότι στην χώρα του ο καθένας πολλά πράγματα έχει κάνει και πολλές επενδύσεις έχουν γίνει για την κινηματογραφική εκπαίδευση. Vision Kino στη Γερμανία, Lyceum Produce Cinema στη Γαλλία, Film Education στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, μερικά, μερικές μόνο από τις πολύ σημαντικές δουλειές που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη αφοσίωση και επιτυχημένα αποτελέσματα. Όμως, δεν θα έπρεπε να κάνουμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Είναι να χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία της κοινοτροφική παιδείας μόνο σε εθελοντική και προαιρετική βάση. Αν πρέπει να προχωρήσουμε σε υποχρεωτική βάση, πρέπει καταρχά να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των δασκάλων. Στη χώρα μου, παραδείγματο χάρη, η εκπαίδευση στα μίντια είναι μόνο μια συμπληρωματική ε, πτυχή των ε, σπουδών του. Ο αριθμός των ταινιών που παράγεται ετησίως στην Ευρώπη διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Από 600, 600 ταινίε σε 1200 περίπου. Όμως, ενώ αυξάνεται ο αριθμό των παραγωγών, ο αριθμός που, των ταινιών που διανέμονται εμπορικά μειώνεται. Και αυτό που μειώνεται πολύ περισσότερο είναι ο αριθμός των ταινιών που ταξιδεύουν και περνάνε σύνορα. Το 2009 το μερίδιο των ευρωπαϊκών ταινιών ε, στην Ευρώπη ήταν 27%. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά για την υπόθεση της Ευρώπης ο αριθμός αυτός είναι παραπλανητικός δυστυχώς γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό του 27% ανήκει στις εθνικές παραγωγές κάθε χώρας. Ένας πολύ μικρός αριθμός, ένας πραγματικά ε, απογοητευτικά ε, μικρός αριθμός ε, ταινιών, ε, ευρωπαϊκών ταινιών ταξιδεύουν στις γειτονικές χώρες. Τα φεστιβάλ έχουν μεγάλη επιτυχία. Ε, Υπάρχουν διάφορα ε, ποσοστά που δείχνουν ε, την επιτυχία αυτή και υπάρχει ε, μια όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για εθνικό ή περιφερειακό περιεχόμενο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Και χάρη στα φτηνά αεροπορικά εισιτήρια όλοι ταξιδεύουμε όλο και περισσότερο. Τα σύνορα ανάμεσα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξαφανιστεί, αλλά οι ταινίε από όλα αυτά τα μέρη στα οποία μας αρέσει να ταξιδεύουμε, ταξιδεύουν όλο και λιγότερο. Αυτή η κίνηση πρόκειται να σταματήσει εντελώς, αν δεν αντιδράσουμε γρήγορα και δεν κάνουμε ε, κάτι σύντομα. Ε, αν δεν κάνουμε κάτι ε, άμεσα, μια ολόκληρη γενιά θα ε, χάσει αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και κοινωνικής διαμεσολάβησης. Χρησιμοποιούμε ξένα εργαλεία από την αλλοδαπή, εισαγόμενα που μας αποξενώνουν ακόμα περισσότερο από την Ήπειρό μας, από τις δικές μας ιστορίες, από τις δικές μας εικόνες, από τις δικές μας γλώσσες. Η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα εξαρτάται από αυτή την ολοκλήρωση. Εξαρτάται από το να μοιραζόμαστε συναισθήματα και κοινέ ιστορίες, όχι μόνο νόμους και χρήματα πρέπει να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας με τις δεξιότητες να αποκωδικοποιούν τις εικόνες, ώστε να ε, επιλέγουν τις δικές μας εικόνες, ώστε να θέλουν η Ευρώπη να ε, παράγει και να προβάλλει την δική της εικόνα, την ταυτότητα προς το μέλλον. Διαφορετικά δεν θα δημιουργηθεί, δεν θα υπάρξει η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Θα υπάρχει και θα απομείνει μόνο η διοίκησή της, έως ότου βαρεθεί τελείως ο κόσμος με αυτή την υπόθεση. Είναι η βαθιά μας πεποίθηση ότι το κύριο καθήκον μας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι να διδάξουμε την αποκωδικοποίηση και την απόλαυση του κινηματογράφου μας και της ιστορίας του. Να καταλάβουμε ε, ε τον ανθρωπισμό του Επομένω, ο ευρωπαϊκό πολιτισμό και η κουλτούρα έχει κάτι το οποίο φέρνει τη διάκριση σε σχέση με τον παγκόσμιο κινηματογράφο ότι ε, συνήθω ε, αφορά κάποιο είδου ε, ιστορίε και συγκρούσει τοπικού περιφερειακού χαρακτήρα είναι κάτι το συγκεκριμένο. Είναι τα, χρώματα, η, κουλτούρα, οι παραδόσει, οι γλώσσε κάθε τόπου. Και έτσι αναδύεται η, πολυμορφία και η πολιτική μου πολυμορφία έτσι μένει ζωντανή. Και η Ευρώπη και η εικόνα της Ευρώπης μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να αντλήσει από μια τέτοια εξέλιξη και αν μπει λοιπόν στην ύλη των σχολείων ο κινηματογράφος έτσι θα μπορέσουμε να ε, του, του ανταποδώσουμε αυτά που χρωστάμε με πολλούς τρόπους και στον κινηματογράφο αυτά που χρωστάμε και στην Ευρώπη και τα οπτικοακουστικά είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και η εικόνα είναι το όπλο του μέλλοντος και σε πάρα πολύ σημαντική συγκυρία κάνετε αυτή την ακρόαση γιατί τώρα σχεδιάζονται οι καθητήρες γραμμές ε, του, του, του, του media και επομένως αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση για το Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει τις ανάγκες του κινηματογράφου και της οπτικοοπτικής βιομηχανίας γενικότερα και αυτό να αντιστοιχεί στις ευρωπαϊκές παγκόσμιες εξελίξεις με νέους τρόπους του να υπάρχει καινούργια προσθεμένη αξία και, και, και καινούργια έσοδα. Το να είναι κανείς για τον κινηματογράφο θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του media στο μέλλον. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα για το καλό της εικόνας της Ευρώπης, για το καλό της ευρωπαϊκής οικονομίας πράγματα τα οποία είναι απόσπαστα συνδεδεμένα. Και αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και γι' αυτό θα πρέπει τα μέλη του Πρεβού Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου να γίνουν οι πρεσβευτέ αυτή τη ενημέρωση για του γηματογράφου ενώπιον κάθε αρχή και εξουσία. και μια που υπάρχει αυτή η νομοθετική τώρα διαδικασία η Ακαδημία μα θέλει να βοηθήσει τα τρία θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να έχουμε μια εκστρατεία για πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία όσον αφορά το κινηματογράφο και το σχολείο. Μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να ξεκινήσει από μια κοινή δήλωση των Προέδρων των Τριών Θεσμικών Οργάνων και από τον ίδιο τον Ζωζή Μανουέλ Μπαρόσο ξέρω ότι υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία 100% το 1999 η Ακαδημία μας ε, προσθέσει για πρώτη φορά τα ευρωπαϊκά Όσκαρ και την ίδια χρονιά ε, η Ευρώπη γιόρτασε τη χρονιά του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Από τότε η Ευρώπη έχει αλλάξει ε, πάρα πολύ και έχει αλλάξει όμως και το οπτικοακουστικό τοπίο. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ένα νέο κινηματογράφο στην Ευρώπη για να μπορέσει να ε, διαμορφώσει την ίδια του την εικόνα ο κινηματογράφος και να είναι αυτό τόσο σοβαρό, τόσο ώστε και τα παιδιά και οι έφηβοι να μπορούν να απολαύσουν και να εκτιμήσουν τον κινηματογράφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Vielen Dank, lieber Wim Wenders. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Wim Wenders. Έχουμε ορισμένου ε, συναδέλφου που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσει, αλλά δεν θα αρχίσουμε την ώρα των ερωτήσεων τώρα. Καταρχήν, θα ακούσουμε μία συνάδελφο σας. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας η Άννα Γιάκερ, που έχει γράψει το βιβλίο European Film Industries και έχει γράψει και πάρα πολλά άρθρα και έχει κάνει ομιλίες για το ΜΕΔΙΑ και την κινηματογραφική πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα Και είναι ε, visiting fellow στο Πανεπιστήμιο στο Bristol, στο University of West England. Και θα μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή συμπαραγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο του Μέντια. Κυρία και έχετε το λόγο. Sorry. Thank you. Co-productions can take many forms and the focus of my talk Για τις κοινωνικές συμπαραγωγές της Ευρώπης θα σας πω. Επί τη βάση επισήμων συμφωνιών α, μεταξύ εμπλεκομένων από διαφορετικά όργανα, φορείς και χώρες. Και κυρίως να μιλήσουμε για πολιτικά θέματα και θέματα πολιτικής ταυτότητας. Η ιστορία της συμπαραγωγής ανάγεται στις αρχές του του κινηματογράφου. Και γι' αυτό έχουν γίνει κάποιε προσπάθειε να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία και αυτό έγινε και με την υπόθεση Film Europe που ξεκίνησε δεκαετία του 20 αλλά δεν πέτυχε γιατί υπήρχε, ήταν πάρα πολύ βάλτος του Παγκοσμίου Πολέμου η βιομηχανία και δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να οργανωθούν και να αντιμετωπίσουν τους Αμερικανούς. Στη μεταπολεμική Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι φορείς ε, κρατικοί οι οποίοι εξασφαλίζουν την κρατική υποστήριξη και βοηθούν πάρα πολύ ούτως ώστε να στήθει στα πόδια της η Εθνική Γυμναστική ε, Βιομηχανία και να συνεργάζονται παραγωγή από διαφορετικές χώρες και η πρώτη τέτοια συμφωνία συμπαραγωγής υπεγράφει μεταξύ Γάλλων και Ιταλών το 1949. Σήμερα ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με τα μειονεκτήματα τέτοιων συμφωνιών, όπως είναι το υψηλό κόστος, η γραφειοκρατία, η ανισότητα μεταξύ των εμπλεκομένων και διάφοροι συμβιβασμοί όσον αφορά τη δημιουργία, τη, τη, τη δαπάνη, το στοιχείο και οπότε έχουμε πάρα πολλές ιστορίες σε σχέση με το πώς γίνονται οι σχετικές ε, επιλογές και αν πληρούνται όλα τα κριτήρια, παρά όλα αυτά όμως μέσα σε πέντε χρόνια ε, βασικά πέτυχε η συνθήκη αυτό το οποίο ήταν ο σκοπός δηλαδή και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι αύξησαν την παραγωγή τους και η απασχόληση επίσης αυξήθηκε και έτσι μπορούσαμε να έχουμε διεθνείς παραγωγές, διεθνή αστέρια και μπορούσαμε αυτά το φιλμ αυτός παντού στην Ευρώπη και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεργασία στα υπάρχοντα πλαίσια που προβλέπει κάθε κράτος μέλος. Βέβαια η Ιταλία και η Γαλλία είχαν κάποια κοινά σημεία, πολιτιστικά, είχαν παρόμοιο σύστημα για κίνητρα και δομή της κοινωνικής βιομηχανίας, αλλά ακόμα και των, των, των φορέων οργάνωσης του κινηματογράφου. Και επίσης υπήρξαν κάποιοι ε, Ιταλοί και Γάλλοι που ήταν ε, αφιερωμένοι στο σκοπό αυτό του να προωθήσουν το ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Παρ' όλα αυτά δείχνουν πάρα πολλές κυρίες κριτικέ, όμω πρόσφατα οι ιστορικοί του του κινηματογράφου άρχισαν να ε, αξιολογούν σαν κάτι πάρα πολύ θετικό εκείνε εξελίξεις και θεώρησαν ότι αυτή η συνεργασία η Ιταλο-Γαλλική έφερε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και για πολιτιστικά ε, και για πλευράς αλλά και κοινωνικής. Οπότε θεωρήθηκε ότι δεν ήταν και τόσο ε, συντηρητικέ συμπραγωγέ όσο τα έργα που προχώρησαν από μία και μόνη χώρα. Τώρα, έχουμε το, το όραμα της Ευρώπης της εικόνας που δεν προχώρησε γιατί πολλές φορές ε, αντίθετα με το ήθελε ο Ζαρμονέ υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές ατζέντε και υπήρχαν άλλωστε τότε και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που βρισκόντουσαν πίσω από το σιδρούν παραπέτασμα. Σήμερα όμως, ε, μετά από 40 χρόνια, γίνονται συνεργασίες, συμπαραγωγές μεταξύ Ευρώπης και του υπόλοιπου του κόσμου. Αντιστοιχεί αυτό στην οικονομική συγκυρία. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει περισσότερες συμπαραγωγές, 47 μέχρι σήμερα, οι δε τις ε, μικρότερες χώρες. Οι περισσότερες ε, ταινίε προέρχονται από συμπαραγωγές. Οι πολυμερείς ε, ρυθμίσεις επίσης από το Media και από το Eurimages έχουν ενθαρρυνθεί και έτσι έχουμε λένε και περισσότερους που εμπλέκονται σε συμπαραγωγές και αυτό ε, μας οδηγεί σε υψηλή κοινοτική παραγωγή στην Ευρώπη από την αρχή της δεκαετίας του 1990. Σε πολλούς τρόπους είναι συναφή αυτά τα οποία προκύπτουν από τις συμπαραγωγές όπως και στις εθνικές παραγωγές. Ε, πάντοτε πρέπει να υπάρχουν κάποιες επιλογές πολιτικές, οικονομικές, νομικές, πολιτιστικές. το Ευρωπαϊκός σχηματογράφο συνοδεύεται από αυτή την πολιτική βούληση να υποστηριχτεί και μέσω της πολιτικής συνεργασίας και ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ε, έχει σχέση με την πολιτική εντολή που είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτές τις ε, παραγωγές που αποδίδουν και αντικατοπτρίζουν τις ε, εικόνες, τη ζωή των Ευρωπαίων, τις μνήμες τα όνειρα, τις πεπιθήσεις, την αναζήτηση ταυτότητας και τα έργα που υποστηρίζονται από το Media και το Your Images είναι παραδείγματα του τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την πολιστική πολυμορφία. Έχουμε επομένως του Αμέλιο, του Χάνεκε, των αδερφών Νταρντέν, ε, τα έργα και και άλλων ε, δημιουργών της Διασποράς, Κότσι, Ζεμουρία, Κίν και όλα αυτά είναι ο κοινό τόπο η πλατφόρμα όπου διερευνάται και διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα ενώ τα ονόματα μεγάλων Ευρωπαίων σκηνοθετών εμφανίζονται ε, να υποστηρίζουν ε, έργα, ε, ονόματα όπως Κεν Λόου, Λας Φοντρία, Άλεν Τάνερ, Κλέντε Λούκα, Λούκας Μπελβόθε, Αγγελόπουλος, Φρίντριχ Θορ, Αντωνιόνι και Βιν Βέντερς, Βόλκερ Σλόντορφ, Μανουέλ Ντεολιέρα, Κισλόφσκι Ζανούσικου, Κουστουρίτσα, Βάιντα, Ιστβαν Σβάμπο, Λουσιάν Φίντιλ, Σαρούνα Σπάρτα, μερικοί μόνο, των οποίων τα ονόματα δεν μπορώ μάλιστα να προφέρω. Τα ταμεία επίση δίνουν μια ε, ευκαιρία σε μια νέα γενιά κινηματογραφιστών να βρουν χρηματοδότηση για τι ταινίε του, ε, ιδιαίτερα, αν όχι αποκλειστικά, στην Ανατολή. Οι ταινίε του έχουν μια ισχυρή ταυτότητα. Έχει μάλιστα υποθεί ότι αποτελούν μία από τις πιο δημιουργικές τάσεις στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Αυτές οι συμπαραγωγές δείχνουν ότι η πολιτιστική ιδιαιτερότητα και η πολιτιστική πολυμορφία δεν είναι πράγματα ασύμβατα μεταξύ τους. Υποστηρίζοντας αυτές τις ταινίες, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βοήθησαν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο να παραμείνει στο προσκήνιο, ε, στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης κουλτούρας. Μια κουλτούρα όπου θέματα πολιτικής ταυτότητας και εκπροσώπησης από την άποψη της εθνότητας, της κοινωνικο-οικονομικής θέσης, της φυλής, του φίλου και της ηλικίας ε, διαρθρώνονται. Δεν είναι μικρό το επίδεγμα αυτό παραγωγή κινηματογραφική στην Ευρώπη σχετίζεται άμεσα με την παρέμβαση τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων στις πολιτιστικές υποθέσεις. Το φιλμ είναι σημαντικό μέσο για την κυκλοφορία του πολιτισμού και είναι επίσης ένα ισχυρό μέσο για την έκφραση της ε, συλλογικής ε, φαντασίας ενός λαού. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι πολύμορφο. Η παγκοσμιοποίηση και η τάση τη ψηφιοποίηση μαζί με τι πρόσφατε εξελίξει στην Ευρώπη επέφεραν ένα κατακαιρματισμό των πολιτισμών καθώ επίση και μια ε, διεθνική προοπτική. Στην ψηφιακή εποχή ο κατακαιρματισμός και η πολυμορφία δεν είναι ένα μειονέκτημα, αλλά η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ποικιλομορφία. Δια κρατικές εξορισμού, οι ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ε, βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Στα ε, τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι έχουν ε, ε, δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ε, ανάπτυξη ε, στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτής της, αυτών των προκλήσεων. Όχι μόνο στη Γαλλία, όπου υπάρχει μια μεγάλη παράδοση και ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενισχύσεων για τις συμπαραγωγές. Αλλά σχεδόν παντού στην Ευρώπη έχουν προκύψει πρωτοβουλίες για τις συμπαραγωγές Πολλές φορές δε, τα αποτελέσματα εμφανίζονται ε, στα διεθνή ε, φεστιβάλ ε, της Ευρώπης, όλο και περισσότερο. Επίσης οι Ευρωπαίοι ε, όλο και πιο πολύ δίνουν τους δεσμούς τους με τις πρώην απικίες τους και δημιουργούν περιφερειακά ταμεία που προωθούν διασυνοριακές συνεργασίες. παρόλο που το οικονομικό κλίμα δεν ευνοεί ε, τέτοιες πρωτοβουλίες διάφορες παραδόσεις ε, συχνά αντικρουόμενες της Ευρώπης ε, όσον αφορά την πρόθεση της πολιτικής πολυμορφίας και η κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κράτη-μέλη σήμερα δεν διευκολύνει το έργο αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις για τον ε, ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Παρ' όλα αυτά, η αναγέννηση εθνικιστικών κινημάτων σήμερα στην Ευρώπη κάνουν πιο επίγουσα την ανάγκη να ε, επιλέξει η Ευρώπη τις πολιτιστικές της ε, προτεραιότητες. Ε, αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι πρώτες ε, γαλλοϊτολικές παραγωγές της δεκαετίας του 50 ήταν λιγότερο συντηρητικέ από τα καθαρά ε, εθνικά ε, φιλμ. Και αυτό ισχύει και για τις σημερινές συμπαραγωγές. Οι ευρωπαϊκές συμπαραγωγές συνδέονται με θέματα ταυτότητας, με τρόπους που δεν θέτουν σε κίνδυνο αναγκαστικά την πολυμορφία των πολιτιστικών συναφιών και των εθνικών και των ευρωπαϊκών. Ε, μπορούν στην καλύτερη περίπτωση όχι μόνο να συμφιλιώσουν, αλλά να συνενώσουν και να εμπλουτίσουν τις ταυτότητες αυτές. Πολλά από τα φιλμ των σκηνοθετών που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι ε, αποτελέσματα συμπαραγωγής ε, με μέσω του ΆΡΤΕ ή προβάλλονται από το ΆΡΤΕ, που είναι ένα ευρωπαϊκό πολιτιστικό κανάλι που προωθεί την ε, ε, πολιτιστική και διεθνή φύση και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Σίγουρα τα κριτήρια αυτά του Άρτε είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σήμερα που είναι τόσο δύσκολο να κάνει κανείς τις επιλογές του. Ε, σε μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οπτικοκουστικού Παρατηρητηρίου ε, περιγράφονται, ε, περιγράφονται οι συμπαραγωγές σαν μια γέφυρα προς την Ευρώπη. δεν είναι καθόλου στενά ευρωπαϊκές συμπαραγωγές, είναι διασυνοριακές και διυπηρωτικές πολλές φορές και ανοίγουν ευκαιρίες και προς τρίτες χώρες να γίνουν εταίρες οι συμπαραγωγές αυτές και έτσι μπορεί να είναι μια γέφυρα και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Σε τελευταία ανάλυση, η κατεύθυνση την οποία θα πάρει ο Ευρωπαϊκός κινηματογράφος εξαρτάται ε, και από τις κρίσιμες επιλογές που θα ληφθούν σε θεσμικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών συμπαραγωγών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάγκερ. Αυτό που μας είπατε δείχνουμε ότι με το πρόγραμμα μας Media και με το Μέτια Μούντος βρισκόμαστε σε σωστό μέσο. Πολλοί από εκείνους που βραβεύτηκαν στα φεστιβάλ έχουν συγχρηματοδοστεί από την Media και ίσως ποτέ δεν θα έχουν μπορέσει να αρθοποδήσουν αν δεν υπήρχε το Media. Λοιπόν, εμείς με τα προγράμματά μας προσπαθούμε πραγματικά να γεφυρώσουμε την Ευρώπη από την Ανατολή προς τη Δύση και από το Βορρά προς τον Νότο αλλά και σε όλο τον κόσμο, όπως το είδαμε με το Media Mundus. Τώρα ακούσαμε τους δύο ομιλητές, θα ήθελα να αρχίσουμε τώρα κάποια συζήτηση. Επτά συνάδελφοι έχουν ήδη ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ κάθε συνάδελφο να μην κάνει δική του παρουσίαση έκθεσης, αλλά να περιοριστεί σε αυτά που δεν έχουν πει οι προηγούμενοι. Ο κ. Μάρτιν είναι ο πρώτος, παρακαλώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέντερς, θα... με ακούσατε παθιασμένο. Με την ανάλυση συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ είμαι πολύ υπερευρωπαίος και συμφωνώ με αυτό που είπατε για την εικόνα που θέλετε να έχουμε. Αλλά είπατε, η δίγηση είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα το media κινηματογράφος θα μπορούσε να είναι ένα μέσο, ένα όπλο. Και αναφερθήκατε στο αμερικανικό όνειρο και στο ευρωπαϊκό όνειρο. Εσείς όμως βλέπετε ότι ο, ο κινηματογράφος ενδυναμώνει την εικόνα του αμερικανικού ονείρου. Εγώ το 1999, μετά από 15 χρόνια ως δημοσιογράφος στους Σπίγελ μπήκα στην πολιτική προωθώντας το ευρωπαϊκό όραμα που βασίζεται στο μενικό ότι όλοι μπορούν δηλαδή, να πετύχουν τα πάντα. Αλλά αυτό είναι μια παγίδα. Υπάρχει μια πραγματική Ευρωπαϊκή ε, Ένωση που βασίζεται στη γραφειοκρατία, στην, ε, στις μεγάλες τράπεζες που σπαταλά τις προσπάθειες σας. Και αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς είναι να γεφυρώσετε από αυτή την πολύ θετική εικόνα που χρειαζόμαστε από κατεπηγόντως για τους νέους. Αλλά δεν πρέπει έτσι να επικαλύψουμε τα προβλήματα. Εν τελευταία αναλύση όλα χρήματα είναι, θα σου πω. Έχω πολλούς φίλους στην κοινογράφο που ήταν εδώ πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό που μας είπαν είναι, αυτός που οριζόμαστε είναι ψηλά. Θέλουμε να μπορούμε στα προ, στα, στους κινηματογράφους να χρη, επιδοτούν οι θέσει των θεατών, στον τόσο αυτές οι υπεροβιές να μπορούν να παρουσιάζονται. Πέρασε ένας χρόνος, δεν έγινε τίποτα. Θα μπορούσε όμως κάτι να γίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η παγίδα των γραφειοκρατών είναι τόσο σημαντική. Την επόμενη εβδομάδα εμείς θα πάμε με 30 άτομα στην Κίνα και όλοι πετάνε ε, business και ε, αντί να πληρώσουν τις 3.000 για το business θέλουν να πληρώσουν 1.200 ορισμένα. Ναι, αλλά θα μπορούσαμε έτσι να απελευθερώσουμε χρήματα για δικά σας σχέδια. Πρόεδρος, παρακαλώ, δεν είναι αυτό το θέμα. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δεν ζητώ τόσο πολύ συγγνώμα. Δεν μπορεί να το αλλάξει ο κύριο Βέντε, ούτε εσεί ούτε εκείνο. Όχι μπορεί γιατί θα μπορέσει να προσπίσει τα θετικά που προσπίσει αλλά και να απαιτήσει τα χρήματα που υπάρχουν στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα 140 δισεκατομμύρια κρυμμένα να τα χρησιμοποιήσουν εκεί που χρειάζεται. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσω αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί και νομίζω ότι οι δύο ομιλητές ο Βιμβέντες και η Άννη Γιάκελ ε, μας είπαν ε, θαυμάσια πράγματα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, γιατί έχουμε κάποιε σημαντικέ αλλαγέ και θεσμικέ μάλιστα να αντιμετωπίσουμε. Από την μια μεριά έχουμε μια συνθήκη που λέει ότι ο πολιτισμό πρέπει να, βρίσκε, να είναι μια διάσταση όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και είναι γεγονό ότι πρέπει να ξαναδώσουμε ψυχή στην εικόνα τη Ευρώπη. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα σημαντικό που είναι η μετατροπή ε, της ε, πραγματικότητας ε, μέσω της οποίας το πολιτιστικό προϊόν μπορεί να είναι ο πρέσβης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά μπορεί να ειδωθεί επίσης σαν μια μεγάλη πρόκληση ε, ε, μιας ε, νέας μορφής πολιτισμού που θα εστίζεται στο πολιτιστικό προϊόν, στην πολιτιστική δημιουργία, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την δημιουργία συμπαραγωγών και για την βιομηχανία τη δημιουργική όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την πράσινη βίβλο της Κομισιόν για την ε, ε, πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία της Κομισιόν και ε, επ' αυτού είχα την ευκαιρία να διαβουλευτώ με τους αρμόδιους στην Ιταλία και δεύτερον, Θέλω να πω το εξή. Αυτό που λέμε για τον αλφαβητισμό των νέων γενεών ε, και τον προβληματισμό που ανέπτυξε ο Βιμ Βέντερ ε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη νέα γενιά είναι μια άλλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τα βραβεία Lux, αλλά τέτοιε προσπάθειε θα πρέπει να τι ενισχύσουμε με πρωτοβουλίε και να επιστήσουμε περισσότερο την προσοχή να προσελκύσουμε τον κόσμο στις πρωτοβουλίες αυτές. Επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική για το θέμα του ψηφιακού χάσματος και της ψηφιακής κουλτούρας. Ε, πρέπει όμως ε, αυτό να το συνδυάσουμε με τον κινηματογραφικό αλφαβητισμό και την ικανότητα ανάγνωσης της εικόνας. Ε, μια άλλη πρόκληση είναι ότι οι ταινίες μας δεν ταξιδεύουν. Δώσατε τα σχετικά στοιχεία. Νομίζω όμως υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά θέματα. Πώς να αντισταθμίσουμε ε, τη μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή που γίνεται στην Ευρώπη ε, ε, για το θέμα του κινηματογράφου του δημιουργού, πώς δηλαδή μπορεί να ανταμυφθεί το έργο του δημιουργού, υπήρξε και ένα σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. πρέπει να το σκεφτούμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό με τη βοήθειά σας για να εξισορροπήσουμε το δικαίωμα του χρήστη, το δικαίωμα ανταμοιβή και αναγνώρισης του δημιουργού και το δικαίωμα βεβαίως των διαφόρων ε, παραγόντων ε, που συμβάλλουν σε μια παραγωγή. Για τον οπτικοακουστικό κλάδο τώρα και την ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία και το μέρος που κατέχει εκεί η ε, ε, δημιουργική βιομηχανία. Είναι ε, ένα 7% του ΑΕΠ. Χρειάζεται μεγαλύτερη επικέντρωση στον πολιτισμό. Και θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς τι προτάσεις μπορούν να γίνουν ή τροποποιήσεις μέσω του προγράμματος Media και του προγράμματος Euro Images αν μιλάμε συνολικά για τον κλάδο κινηματογράφος και οπτικοακουστικά ε, ή χωρίζονται οι δύο κλάδοι και τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προωθηθούν οι συμπαραγωγέ, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι και τόσο εθαρρυντική όσον αφορά τι συμπαραγωγέ. Και επίση έχουμε δεσμευτεί να ζητήσουμε να υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης των κρατών μελών στην ε, ψηφιοποίηση, σε, κονδύλια μάλλον, για την ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών ε, αιθουσών γιατί σήμερα αυτό γίνεται μόνο το κατά παρέκκληση και με κρατικές ενισχύσεις. Λέω λοιπόν ότι η ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αιθουσών ε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταγωνιστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Monsieur Cavada, s'il vous plaît. Ο Καβαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τεράστια ευτυχία να σας ακούμε και να άπτεστε της πραγματικότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αναφέρομαι σε εσά, ε, κυρία μου, αλλά και σε αυτά που είπε και ο κύριος Βιβέντος, φυσικά. Ο ιστορικός είπε ότι οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους ε, εκτίθενται στον κίνδυνο να την ξαναζήσουν. Δεν τους ακούσαμε και αρχίζουμε να ξαναζούμε μια ιστορία, ε, ιστορία που κατέρευσε την Ευρώπη. Βλέπουμε τι φτάνει προς την εξουσία. Σε ορισμένες δύο χώρες είναι ήδη οι άνθρωποι αυτοί εκείνοι που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και αυτό σκοπίζεται σαν οξύ σε, ένα, σε ένα νηστό ένα εθνικιστικό ε, αίσθημα και όχι ευρωπαϊκό. Αν ήμουν επεσέδωση θα έλεγα ότι αποτύχαμε. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε το ευρωπαϊκό αίσθημα που χρειαζόμαστε γιατί οι τεχνοκράτες και εκείνοι που φοβούνται εύκολα είπανε προς τους υπεύθυνους εξουσίας ότι το αίσθημα το να ανοίγει κανένα στην Ευρώπη είναι αντίθετο, είναι αρνητικό για το εθνικό συνέστημα. Γι' αυτό ε, επικροτώ απόλυτα τον κύριο Βέντερς και το αποδεικνύει και το έργο σας. Υπάρχουν δύο-τρία σημεία που θίξατε και εσείς κυρία μου. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα έργο χωρίς ε, οικονομικούς πόρους και ο πολιτισμό είναι ένα κλάδο τη οικονομία. Αν δεν υπάρχουν χρήματα δεν θα υπάρχει δημιουργία, δεν θα υπάρχει επικοινωνία και διάδοση των ε, έργων αυτών. Πριν από 20 χρόνια έπεσε το τείχο του Βερολίνου, αλλά εκεί εμεί που ζούμε στη Δύση γνωρίζουμε πραγματικά του λαού που είναι τώρα πια σύμμαχοί μα, που είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα έργα που μα παρουσιάζουν τα δράματα που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί την εποχή που εμεί. Ε, έτσι καναμερολογίες, δεν κοστίζει και τίποτα. Υπάρχουν μεγάλα σημαντικά έργα που ήρθαν την Κεντρική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, αλλά δεν είναι αυτά επαρκή. Εγώ είμαι Ευρωπαίος από τη Γαλλία. Εάν κάποιον Γάλλο ρωτήσετε έτσι, τι έγινε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ουγγαρία παραδείγματος χάρη, δεν θα σας πει πολλά. Φτάνω σε δύο προτάσεις που τονίσατε εσείς που θα πρέπει να προσπίσουμε κύριε Βέντες κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες χώρες, η δική μου λειτουργήσε καλά νομίζω εδώ, πρέπει να βρούμε ένα σύστημα χρηματοδότησης της δημιουργίας, όχι μόνο για τον κινηματογράφο, η πρόεδρος το ξέρει, και για τη δημιουργία των οπτικοστικών στην τηλεόραση φυσικά. Δεν θεωρώ δημιουργία από το 20 αυτά που βλέπαμε, βλέπουμε στα κανάλια μεγάλη κατανάλωσης. Αυτά πάνε χρηματοδοτούνται από την διαφήμιση, εντάξει. Αλλά <clears throat> πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι θέλει να αναπτύξει την, τον πολιτισμό και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτελέσει το έργο της. Δεν το έχει κάνει ακόμα θα πρέπει εκτός από τα εθνικά ταμεία να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό ταμείο για τη δημιουργία αλλά ακόμη και τη μετάφραση έργων σε εθνική ψηφιακή μορφή. Αλλά δεν πρέπει να τους δώσουμε μόνο ψυχία. Είναι επικίνδυνο αν δεν χρηματοδοτήσουμε σωστά. Ε, δεύτερο, και μπορώ να σας δώσω δίκαιο εδώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βέντελς, θα πρέπει να φροντίσουμε η έννοια αυτών των εργών να διδάσκεται στα παιδιά για να μπορούν να ωφεληθούν από τις εικόνες αυτές, να είναι θύματα απλώς. Πραγματικά. Σε ένα σώμα που δισκάζει για το μέλλον της Ευρώπης, ε, χαίρομαι να ακούσω αυτά που άκουσα και που μας είπατε. Πρώτα, ευχαριστώ κύριε Καβατά. Ο κύριος Σκουρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική σήμερα ημέρα για το κοινοβουλίο μας, χάρη στις παρεμβάσεις των δύο φιλοξενούμενών μας. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να μιλάμε για την Ευρώπη ε, σαν ψυχή, σαν όνειρο, σαν συνέστημα, σαν ταυτότητα. Ακούσαμε ε, μια προφητική σχεδόν ε, ομιλία για μια μελλοντική ε, αντίληψη της Ευρώπης που μερικές φορές λείπει από αυτές τις αίθουσες. Όλα τα μέτρα αυτής της ε, Επιτροπής, ξεκινώντας από την πρόεδρό μας, προσπαθούν να μοιήσουν τους άλλους συναδέλφους σχετικά με την σπουδαιότητα του πολιτισμού και του τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε ε, να, έχουμε μια, να δούμε μια Ευρώπη ε, διαφορετική από αυτή ε, που γίνεται συνήθως αντιληπτή σαν μια αντιπαθητική γραφειοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα είναι σημαντική η ημέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κάτι πολύ απλό στους ε, καλεσμένους μας. Ένα πράγμα πολύ απλό. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν κοινοβούλιο για να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην πραγματοποίηση αυτού του ονείρου. Ξέροντας ότι η περίοδος δεν είναι πολύ ανθυρή από οικονομικής απόψεως. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. Σαντιάγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μία συγκεκριμένη στον κύριο Βέντρε. Μα είπατε κάποια αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά το τι γίνεται με τι ευρωπαϊκέ ταινίε σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, Επομένω, ε, ε, το ίδιο γίνεται και με πολλού από εμά που όταν πάμε σε κάποιε άλλε πόλει βλέπουμε κάποια έργα που θα θέλουμε να δούμε, αλλά όταν γυρίζουμε στη δική μα πόλη δεν παίζονται για να δούμε αυτά τα έργα. Εγώ θέλω την ελεύθερη αγορά, δεν θέλω να μου επιβάλλουν τίποτα. Όμω, τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα τόσο ώστε να διευκολύνουμε ένα σωρό Ευρωπαίου που θέλουμε να δούμε ευρωπαϊκό κινηματογράφο που μα αρέσει. Η ε, πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριο Μπελέτ. Ε, Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Βέντας για την πανευρωπαϊκή πρόταση για την κρεματογραφική παιδεία των παιδιών. Είμαστε μια επιτροπή πολιτισμού, εδώ θα πρέπει να το υποστηρίξουμε απόλυτα. Ε, είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν οι ε, και οι πολίτες του μέλλοντος να έχουν πρόσβαση στην κοινή μας αυτή κληρονομιά. Η πρόεδρος μας, η κυρία ΠΑΚ θα πρέπει να έρθει σε επαφή νομίζω με τους εθνικούς περιφερειακούς συναδέλφους σας για να ξεκινήσει η πρωτοβουλία αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσον στο πρόγραμμα Μέντια υπάρχει δυνατότητα υποστήριξη ή θα πρέπει να έχουμε από αλλού την υποστήριξη αυτή τη πρωτοβουλία. Δεν είναι θέμα χρημάτων νομίζω, είναι θέμα πολιτική βούληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω. Έχω ένα σημαντικό ερώτημα προς τον κύριο Βέντες. Όταν μιλάμε για την πρωτοβουλία αυτή, που μιλάμε... μιλάμε... What are we talking about? Is it not... Is the, is the game... Ε, ε, μιλάμε και για τη δημιουργία των παιχνιδιών. Ε, είναι και αυτό ένα τμήμα της εβδόμης τέχνης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω ουγγρικά. Αγαπητέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας ακούμε, να μας τα λέτε και το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και συγκεκριμένα για τους νέους. Θα δείτε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πόσοι νέοι ενδιαφέρονται για, ε, για τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Και επίσης ε, θα πρέπει να τα υπόψη το πόσο δυνατό είναι ο κινηματογράφο, μια που και το αμερικανικό όνειρο είχε σαν θεμέλια και τον αμερικανικό κινηματογράφο. Όμω και εμεί επομένω θα πρέπει να δούμε πώ ο κινηματογράφο θα βοηθήσει το ευρωπαϊκό όραμα. Και βλέπουμε ότι το 80% του, του, του υλικού, του πολιστικού είναι ε, προερχόμενο προέρχεται από την ε, Αμερική. Βλέπουμε ότι υπάρχει λοιπόν μια πολιτιστική εισβολή, φυσικά ξερώντα τα κλασικά έργα. Και γι' αυτό και θα πρέπει να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής παραγωγής, των ε, Κουστουρίτσα, τον Αλμοδόβαρ, γιατί Όλοι αυτοί οι δημιουργοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αναβάθμιση, την προώθηση του ευρωπαϊκού οράματο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επίση να γεφυρώσουμε κάπως αυτό το χάσμα το οποίο λένε και μεγαλώνει μεταξύ Ευρώπη και νέων. Αυτή η στρατηγική Youth on the Move, η στρατηγική για το 2020, όλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουμε το χάσμα αυτό μεταξύ νέων και Ευρώπης και το Κοινοβούλιο επίσης μπορεί να βοηθήσει και για τους ε, τσιγκάνους ε, έχουμε στρατηγικές ε, και επομένως αξίζει όλα αυτά να περάσουν μέσα από μια στατική για τον κινηματογράφο. Και αυτός ο κλάδος, αυτή η βιομηχανία θα πρέπει να δεχθούμε το πόσο προωθεί πολιτιστικές ε, αξίες. Και αυτό θα πρέπει να κάνει και θα, θα πρέπει να καταλήγει να γίνει mainstream, να γίνει ένα εμπορικό προϊόν και έτσι να φροντίζει μόνο να παραγάγει κάποια έργα τα οποία να είναι απλώς εύκολα. Βλέπουμε ότι πρόκειται επομένω για δίκοπο μαχαίρι, ε, γιατί θέλουμε κυρίως να έχουμε αισθητικές αξίες που να, να, να, να προωθούνται, γιατί ξέρετε ακόμα και τα κινούμενα σχέδια είναι χρήσιμα για τους μικρούς, αλλά ο κλάδος των κινούμενων σχεδίων, εκεί και εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εισβολή αμερικανική. Εμεί στη χώρα μου την Ουγγαρία έχουμε μεγάλη παράδοση, Όμω θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την αμερικανική εισβολή. Τελειώνω, τελειώνω πρόεδρε, σε ένα λεφτάκι. Γιατί έλεγα ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ε, παλιότερα οι καινούργιες ήταν πάρα πολύ μικρέ και τώρα είναι multiplex, ε, έχουμε ολόκληρα εμπορικά κέντρα με τα multiplex και όπως στην Αμερική. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε μια στρατηγική αυτή να αποτυπωθεί με μολύβι και χαρτί και επίσης να έχουμε και στέρεη οικονομική βάση, αρκετούς πόρους. Αν αυτό το, το κάνουμε θα πετύχουμε στο στόχο μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις εξαιρετικές αυτές ε, παρουσιάσεις ε, που ευνεούν όλους μας. Ε, εγώ ε, ενδιαφέρομαι για, ε, για τον κλασικό πολιτισμό και θα ήθελα να αναφερθώ στον βυζαντινό πολιτισμό που έζησε για πάνω από χίλια χρόνια και τον πανσλαβικό ε, πολιτισμό. Και εκεί η εικόνα είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. στον βυζαντινό κόσμο η, εικόνα του κόσμου ήταν η εικονογραφία που μετέφερε ιδεολογίες και συναισθήματα και μετά τον 14ο, 15ο αιώνα στη Μόσχα και στο Κίεβο ο Αντρέι Λιούβο ε, έδωσε την σλαβική ψυχή μέσα από τις εικόνες. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν εσείς βλέπετε αυτή τη σύνδεση με την ιστορία δεν ζούμε πλέον σε έναν ε, ε θρησκευτικό κόσμο, δεν έχουμε μία ε, και μόνο θρησκεία. Ο κόσμος όμως ε, είναι ιερός. Δεν μπορούμε να έχουμε την Ευρώπη χωρίς έναν ανθρώπινο όν που αισθάνεται, που σκέφτεται, που γεννιέται και πεθαίνει. Γι' αυτό με συγκίνησαν τόσο πολύ οι παρουσιάσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Σας ευχαριστώ κύριε Βεντός για τα τόσο καλά που μας είπατε που τονίσατε ποια είναι η σημασία του κινηματογράφου για την κοινωνία και μέσα στην κοινωνία. Ιδίως αυτό που είπατε όσον αφορά την ε, ε διεύρυνση των ε, ικανοτήτων για τα διάφορα μέσα να διευρυνθεί για να καλύψει και τον κινηματογράφο στα πέδια της ε, εκπαίδευσης των παιδιών, αυτό μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Και πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά στα κράτη-μέλη να γίνει αποδεκτό ότι αυτό θα πρέπει να περάσει ίσως στη δεκταία ύλη των σχολείων και θα πρέπει να δούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε συμπραγματικά Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε για το πώς μπορεί να βοηθήσει ο κινηματογράφος στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αυτά που είπατε ήταν πολύ σωστά. Από την άλλη μεριά πιστεύω ότι εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα με τον κινηματογράφο, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο κινηματογράφος, αυτή η ταινία θα πρέπει να είναι ελκυστική για πάρα πολλούς ανθρώπους για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η ταυτότητα. Και βέβαια το ότι αρέσει σε πάρα πολλούς δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το αμερικανικό mainstream του Ναντίο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο πόσο ελκυστική είναι μια ταινία και στο ε, ε, πόσο υψηλή ποιότητα είναι. αλλά θα πρέπει νομίζω να πετύχουμε την ελκυστικότητα για το κοινό που έχουν οι Αμερικανικέ νέε. Και γι' αυτό σα ρωτάω και του δύο, και τον κύριο Βέντε και την κυρία Γέγκα. Και τι πιστεύετε ότι εμεί ω πολιτικοί μπορούμε να κάνουμε, εκτό από τα χρήματα που πάντα βέβαια προσπαθούμε να διαθέσουμε περισσότερα από ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα Μέντια ή οπουδήποτε αλλού. Πέρα από τα χρήματα, τι μπορούμε να κάνουμε, ούτω ώστε να προωθήσουμε αυτή την ιδέα της, Αμερικαν... της ε, ευρωπαϊκής ε, κινηματογραφικής ταινία που έχει πραγματικά αυτή την ελκυστικότητα για τους πολίτες, για το ευρύ κοινό. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βοηθήσουμε περαιτέρω τους Ευρωπαίοι πολιτικοί. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση. Μετά έχουμε άλλη μια δυνατότητα για να ερωτήσεων. Τώρα ζήτησαν και άλλοι δύο το λόγο, αλλά ίσως θα μπορέσετε εσείς να μιλήσετε στον επόμενο γύρο. Δείξτε παρακαλώ κατανόηση. Αλλιώ οι άλλοι ομιλητέ δεν θα μιλήσουν. Θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα καταρχήν στον Βιμβέντε να απαντήσει στι ερωτήσει αν θέλει. Παρακαλώ. Such a Τόσες ερωτήσεις. Και όταν σα άκουσα να βάλετε αυτές τι ερωτήσεις, συνειδητοποίησα ότι είμαι αισιόδοξο. Ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ταξιδεύω πολύ. Παντού στον κόσμο. Πραγματικά ταξιδεύω πολύ. Οπότε μπορώ να διαπιστώσω πόσο σεβασμός χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο προ την Ευρώπη και για τον κινηματογράφη της. Βεβαίω όλοι θεωρούν την οικονομική ε, δύναμη η Ευρώπη, αλλά κυρίως τη σέβονται για τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα της και και για τον κινηματογράφο της. Όμως αυτός ο σεβασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μακάρι να μπορούσα να σας ε, το εκφράσω το πόσο θα ήθελα η Ευρώπη να μπορεί να αντικατοπτρήσει τη, δική της εικόνα προς τους δικούς της πολίτες σε σχέση με αυτόν τον σεβασμό προς τον πολιτισμό και έτσι να μπορούσε αυτό το ατού να το χρησιμοποιήσει η Ευρώπη γιατί αυτό το πλανήθημα το έχει η Ευρώπη, το ξέρουν όλοι οι άλλοι και το ξέρει η Ευρώπη. παρά το έλλειμμα επομένως να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς ε, πολιτισμό και χωρίς ε, κινηματογράφο θα είχαμε εξαφανιστεί από το χάρτη. Ε, άρα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι όχι να απαντήσω όλες τις ερωτήσει ερωτήσεις το πώς και τι θα γίνει για το κάθε σημείο αλλά απλώς θέλω να προβληματιστούμε για το μέλλον, το, το, τους μέλλοντες θεατές, ακροατήρια, το τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλιστεί η σχετική κοινογραφική παιδεία. Γιατί αυτό χρειάζεται για το μέλλον. Αυτοσεβασμός. Βελτίωση της εικόνας της Ευρώπης προς την ίδια. Μιλήσαμε για την ψηφιοποίηση, πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Ακριβώς σαν το copyright. Τα πνευματικά δικαιώματα και στα πλαίσια αυτής της ε, συζήτησης όσον αφορά την ε, ψηφιοποίηση παρακαλώ συνέχεια να έχετε υπόψη το ότι χρειάζεται να ψηφιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερε οθόνε στην Ευρώπη και αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φρενάρουμε την προσβασιμότητα στον κινηματογράφο να μην υπάρχει κωδικοποίηση να μην περιορίζεται η πρόσβαση στον κινηματογράφο και, και του κινηματογράφου στην διανομή, αλλά να βοηθιέται αυτή η διανομή. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους κινηματογράφους οι οποίοι δίνουν ε, πιο σκληρή μάχη, γιατί πάρα πολλές φορές ε, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται, δεν έχει κανείς τα χρήματα για την ψηφιοποίηση. Κάτι είναι με σταυρωμένα χέρια και παρακολουθεί τι γίνεται στον υπόλοιπο χρόνο, στον υπόλοιπο κόσμο. Συγγνώμη. Άρα να πρέπει να δώσουμε χείρα βοηθεία, αλλά αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο που οι ψηφιακέ οθόνε να μην είναι κάτι το περιορισμένο. Και να μπορούν τα δικά μας προϊόντα και οι δικές μας ταινίες να προβληθούν εκεί. Πολύ σημαντικά. Αυτό λέω για το μέλλον και επίσης βλέπουμε ε, τι γίνεται με τη βιομηχανία του παιχνιδιού, ε, πόσες ταινίες προέρχονται από τέτοια ε, computer games. Βεβαίω και είναι σημαντικό να διδάξει κανείς τα παιδιά τι γίνεται με τα παιχνίδια αυτά για υπολογιστέ. Πώς κανείς μπορεί να συνεπάρξει με αυτά τα παιχνίδια, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν βοήθεια μόνο από τους γονείς ίσως. Αλλά κανείς δεν τα βοηθάει. Για αυτό πώς να το πούμε. Πώς το να αυτή την εξάρτηση. Γιατί έχω δει παιδιά που κατά τα άλλα είναι υπέροχα και έχουν φαντασία να εκδηλώνουν τέτοια εξάρτηση. Να επομένως ακόμα ένα στόχος της εκπαίδευσης της παιδείας. Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις φαντάζομαι πιέζει ο χρόνος. Εσείς κυρία Γέγελ. Δύο λόγια μόνο. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να οργανώσουμε κάτι που να είναι μια γιορτή για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Μια γιορτή, ένας γιορτασμός ε, της ποικιλία που υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Είναι κάτι που λείπει νομίζω. Δεν γιορτάζουμε το πράγμα αυτό στην Ευρώπη. Και να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Βέντερς. Ε, οι άλλοι λαοί σέβονται τον πολιτισμό μας, τον θαυμάζουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντοτε το βρίσκω ε, ε, βρίσκω ότι γίνεται κάτι πολύ περίεργο. Αν μια ταινία είχε επιτυχία στι Ηνωμένε Πολιτείε, πάνε και την βλέπουν ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι. γιατί? Και οι Αμερικάνοι δοξάζουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και πολλοί άλλοι λαοί, πολλές άλλες χώρες. Γιατί, λοιπόν, να ε, ε, μην το κάνουμε κι εμείς αυτό. Δεν είμαστε καλοί στο να τιμάμε το δικό μας κινηματογράφο. Τώρα, ε, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αν μπορεί να προωθήσει το ευρωπαϊκό όνειρο, αυτό είναι ένα πιο δύσκολο ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερη χρήση του ίντερνετ. Των νέων ε, μέσων, των μέσω δυνατοτήτων που προσφέρονται και που μπορούν να οργανώσουν μια συζήτηση μέσω ε, δικτύων. Είτε πρόκειται για τον κινηματογράφο, είτε για να μάθει κανείς ε, τι γίνεται σε σχέση με τον κινηματογράφο. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στους δύο επόμενους ομιλητές. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόμαν Γκούτεκ, ο οποίος είναι ιδρυτής ε, ε, μια από τις πιο σημαντικές από ποσοτική και ποιοτική άποψη ε, διανομής στην Πολωνία. Νομίζω ότι είναι ένας ήρωας της προώθησης των ελληνικών ταινιών σε μια αγορά που όταν ξεκίνησε ήταν ε, μονοπόλιο. Ε, και θα μας μιλήσει σήμερα για το εξής. Θα μπορείτε να το φανταστείτε καν. Ότι οργανώνει στο Βάτσλαβ το πρώτο ε, ανεξάρτητο αμερικάνικο φεστιβάλ μετά ε, από το πρώτο φεστιβάλ ρωσικού κινηματογράφου που οργάνωσε. Έχετε το λόγο. Polish, it's uh, θα μιλήσω πολωνικά. Ε, γιατί οργανώνω ε, στο Βρότσβο στη Βρεσλάβια ε, ένα φεστιβάλ αμερικάνικου κινηματογράφου που ξεκίνησε την Κυριακή και κράτησε πέντε μέρες. Οργανώσαμε αυτό το φεστιβάλ για να ε, δώσουμε νέα ζωή ε, σε αυτή την εικόνα του Αμερικανικού κινηματογράφου που σχετίζεται περισσότερο, είχε σχετιστεί με το popcorn. Θέλαμε να δείξουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο του Αμερικανικού κινηματογράφου. Ότι υπάρχει και ο ανεξάρτητος Αμερικανός κινηματογράφος και επομένως να δείξουμε και κάποιες κλασικές ταινίες, οι μισές σχεδόν ήταν τέτοιες όπως το Καζαμπλάνκα, όπως το Πολίτης Κέιν και πολλές άλλες. Ήρθανε μαθητές στον Ρόδα Σχολεία από την Βαρσοβία, ε, ήρθανε, αγοράστηκαν εισιτήρια και συζητήσαμε για όλα αυτά. Εγώ πρεσβεύω την πολυμορφία και ε, θέλω να υπάρχει προσβασιμότητα της το, το, το κινηματογράφο, τον Αμερικανικό, αλλά φυσικά και τον πολιτικό κινηματογράφο. 16 χρόνια εγώ ε, ασχολούμαι με αυτο τον φορέα μας. Ε, ε, έχουμε προβάλει 300 ταινίες, περισσότερες είναι ευρωπαϊκές και είχαμε περίπου 10 εκατομμύρια που ήρθαν για να παρακολουθήσουν αυτές τις ταινίες. Νομίζω ότι είναι ένας αριθμός εντυπωσιακός, οπότε και αυτό νομίζω καλύπτει αυτό το οποίο ερώτησε η κυρία Πρόεδρος. Ελπίζω σας καλύπτω κυρία Πρόεδρε. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι βλέπω εκατοντάδες ταινίες κάθε χρόνο σε φεστιβάλ παντού. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πολυμορφία, ακόμα εξελίσσεται, μεγαλώνει, αλλάζει ο κινηματογράφος. Μπορεί να μας εκπλήξει στην Ευρώπη και ε, έχουμε το θέμα του πώς θα φτάσουμε στον θεατή γιατί μπορώ να σας πω τι γίνεται για τα έργα τα οποία εμένα μου αρέσουν δηλαδή αυτά που έχουν κάποιοι νέοι, κάποιοι ανεξάρτητοι που προέρχονται από μικρές χώρες και αυτοί δυσκολεύονται να ε, τους μάθει ο, ο γιατί τα πράγματα έχω αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη 20 30 γιατί τότε το ευρωπαϊκό σινεμά ήταν κάτι πολύ πιο προβεβλημένο και το είχαμε Ρότερνταμ, Κα, τις Κάνες, τη Βενετία, αυτά τα φεστιβάλ, εκεί κανείς αν πάει μπορεί να διαπιστώσει την πολυμορφία, τον πλούτο του κινηματογράφου στην Ευρώπη, όμως τώρα ε, περνάμε μια εποχή μετασχηματισμού, το παλιό αναλογικό ε, πρότυπο, Τώρα περνάει μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση, οπότε και εμείς οι επαγγελματίες, ε, οι διανομείς, οι, όλοι οι ασχολούμενοι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνήθειες, τα νέα γούστα του κοινού, θέλουν προσβασιμότητα κατά παραγγελία, on demand, ακριβώς όπως γίνεται και με το ίντερνετ και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να συνδυάζει τις ανάγκες του θεατή και ταυτόχρονα να έχουμε κάποιο πρότυπο ε, επαγγελματικό και έτσι να είναι δυνατόν οι εταιρείε να επιβιώσουν, να, να παραγάγουν τις ταινίε τους και έτσι να προκύψει φυσικά και εισόδημα για τους ε, παραγωγούς. Πάντως για τις ευρωπαϊκές ταινίες θα πάντα είναι εύκολα, ο κύριος ε, Βέντερς μας τα είπε μας εξήγησε ότι το μερίδιο στην αγορά των ευρωπαϊκών ταινιών δεν είναι αρκετό. Και οι διανομής συχνά δυσκολεύονται πάρα πολύ να μπορέσουν να βγάλουν κάποιο κέρδος από την διανομή όσον αφορά κάποιες ξένες ταινίες Υπάρχουν και τα σχετικά έξοδα για την αδειοδότηση. Βεβαίως υπάρχει κάποιο εισόδημα που προέρχεται από κάποιες παραδοσιακές μορφές χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων όπως από την πώληση των ε, δίσκων. Βεβαίως το εδώ είναι και το θέμα της ε, παράνομης ε, του παράνομου κατεβάσματος ταινιών από το διαδίκτυο θα πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται και σε σχέση με τα κρατικά κανάλια, γιατί εμείς ε, δεν καταφέραμε να πείσουμε τους, τα κρατικά κανάλια στη, στην Πολωνία να δείξουν τις ταινίες μας. Προσπαθούν τα κρατικά κανάλια στην Πολωνία να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά και άρα το θέμα δεν είναι μόνο ο συναγωνισμός με τους Αμερικανούς αλλά το θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα καταπολεμηθεί αυτή η τεράστια πειρατεία. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Χηματογράφο να ανταγωνιστεί τα παιχνίδια που παίζονται σε υπολογιστή είναι όλο ένα και πιο ελκυστικά και πιο περίπλοκα. Ε, έχουμε και όλες, όλα αυτά τα σύριαλ που είναι έτσι ακριβά, ε, εντυπωσιακά. Και έφτασε ο Ευρωπαϊκό Κινηματογράφος να στοχεύει μόνο σε κάποια Elite. Έτσι όπως είναι αυτή η κατάσταση βεβαίως και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να εξασφαλίσουμε ε, αυτού του είδους την, την κουλτούρα του κινηματογράφου που να, να περάσει μέσα από την ύλη του σχολείου. Να μάθουν τα παιδιά, να, να μάθουν και οι μεγάλοι για, την παράδοση αυτή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Θα πρέπει να καλυφθούν ε, νέες παραγωγές αλλά και τα κλασικά έργα. Ένα σωρό παραδείγματα τοπικά έχουμε, πάντως εγώ θέλω να υπάρχουν κάποιες ε, συστημικές λύσεις. Έχουμε τους νέους ορίζοντες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Καλύπτει 50.000 ανήλικους και νέους από ένα σωρό πόλεις και πάνε στο σινεμά μια φορά το μήνα μετά συζητούν για την ταινία. Πολλές φορές μιλούν με τον δημιουργό της ταινίας και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μια φορά. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα και καλύπτει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε, όλη της, σε τη διάρκεια. Δεν έχω τώρα χρόνο να σας πω τις λεπτομέρειες του προγράμματος, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και κατά το θερινό μας φεστιβάλ στο Βρότσλαφ έχουμε 200 δάσκαλους οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορα εργαστήρια, έχουμε πολλούς θεατές και έτσι προσπαθούμε να περάσουμε την υπόθεση και μετογράφους στο σχολείο και αυτή είναι πολύ σημαντικό το ότι φέρνουν μαζί τους μαθητές τους. γιατί πολλές φορές οι γονεί δεν μπορούν να αφήσουν κάποιον 16χρονο να πάει μόνος του σε ένα κοινοδό φεστιβάλ σε μια άλλη πόλη. Όταν όμως συνοδεύει ο δάσκαλος, αυτό γίνεται. Και το Πολωνικό Ινστιτούτο του Κινηματογράφου έχει αγοράσει τα σχετικά δικαιώματα και τα έχει διανύμει όσον αφορά τις ταινίες τις, ε, και του μικρού μήκους και έχουμε 15 πακέτα όσον αφορά τα κλασικά πολωνικά έργα, τα στέλνουμε σε σχολεία με μπροσούρες σε σχέση με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ταινίες για τη γλώσσα, για την ιστορία, για την ιστορία της τέχνης. Είναι πρωτοβουλία εύκολη σχετικά, εάν αυτό αφορά πολωνικές ταινίες. Βέβαια για το διεθνή κινηματογράφο τα πράγματα περιπλέκονται. Είναι θέμα βέβαια εφαρμογής. Και έτσι θεωρούμε ότι προάγουμε τον πώς θα περάσει ο κινηματογράφο στα, στα παιδιά μου, στα εταιρεία. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στη Βαρσοβία, πάνω στο, στο κινηματογράφο μου και βλέπουν στην μεγάλη οθόνη το έργο, τους αρέσει, και γι' αυτό θεωρώ ότι όταν μεγαλώσουν θα ξανάρθουν. Βέβαια και το διαδίκτυο βοηθάει. Και θα έπρεπε να υπάρχουν ψηφιακές βιβλιοθήκες ε, στο ίντερνετ και έτσι να είναι πιο εύκολη η προσβασιμότητα ή στι κλασικέ ταινίες, θέλει κανεί να βρει τον Μπρούστον Ντοστογεύσκη, μπορεί να το κάνει. Θα έπρεπε το ίδιο να γίνεται αν θέλει να ψάξει μια ταινία του ή του Αντωνιόνιου. Όλοι βέβαια βλέπουμε στο Ιντερνετ κάποιε ταινίε και πολλέ φορέ κατεβάζουμε παράνομα ταινίε, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την νόμιμη πρόσβαση. Πού να βρει κανεί εύκολα τώρα και νόμιμα ένα έργο για τσιγκάνους. Θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Έχουμε τα ευρωπαϊκά Όσκαρ, είπαμε, ε, έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και 20 χρόνια έχουμε το διαγωνισμό και το βραβείο Λουξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Λουξ. Είναι κάτι που θα βοηθήσει νομίζω. Κάποιες ταινίες. Κάποιες ταινίες που προβάλλονται παντού στην Ευρώπη. Είναι σημαντική η υποστήριξη. και κάποιους άλλους φορείς ε, που έχουμε, κάποια δίκτυα διανομής. Όμως θα πρέπει να βρεθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο βιώσιμο, να βοηθηθούν αυτές οι εταιρείε. Να μπορέσουν αυτές οι εταιρείε να λειτουργήσουν υπό την σημερινή συγκυρία. Και η χρηματοδότηση της διανομής με το πρόγραμμα Media ίσως είναι το κλειδί. Είναι ένα πετυχημένο μέτρο επικούρησης του σινεμά. Λειτουργεί εύρυθμα. Γιατί χωρίς τη βοήθεια του μίντια πάρα πολλά δεν θα είχαν ποτέ διανεμηθεί. Πάντως, παρά την ύπαρξη του προγράμματος, πάρα πολλέ ταινίε. Τελικά δεν φτάνουν στις αίθουσε, μας τα είπε ο κύριος Βέντερς. Έχουμε ε, χίλιες, χίλιες ταινίες που παράγονται στην Ευρώπη αλλά οι μισές από αυτές δεν φτάνουν ποτέ στις αίθουσες. Είδε. συγχρηματοδότηση, για κλπ. Όλα αυτά δεν έχουν νόημα εάν μια ταινία δεν φτάνει στις αίθουσες. Βέβαια, ακόμα και αν προβάλλονται τελικά σε κάποια αίθουσα, αυτό κρατάει μόνο καμιά εβδομαδούλα δεν έχουν οι μικροί διανομής αρκετά χρήματα για να κάνουν αυτό που πρέπει. Άρα για μας τελικά μετράει η φήμη, καλή κουβέντα που θα πει ο ένας θεατής τον άλλο. Πιο πολλές φορές λοιπόν κάποιος ξέρει για μια καλή ταινία, θέλει να πάει να το δει, αλλά δεν παίζεται πια και δεν μπορεί να τη δει την ταινία. Ας πούμε, η εταιρεία μας αγόρασε τα δικαιώματα για ένα γερμανικό έργο την Grosse Stille» τρίωρο έργο, σχεδόν χωρίς διαλόγους και είχαμε στην αρχή τρεις κόπιες του έργου. Μου άρεσε το έργο και ήμουν σίγουρος ότι θα αρέσει και στον κόσμο στην Πολωνία. ξεκινήσαμε στον κινηματογράφο Μουράνο, μια κόπια και ήταν φοβερές οι ώρες του κόσμου περίμενε για να το δει και σε άλλες ταινίες για άλλες κόπιες πήγαν ε, και έξι μήνες το δείχναμε και είχαμε τελικά 50.000 Πολωνών που πήγαν να δουν το έργο αυτό. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί θέλω να πω ότι χρειάζονται αίθουσε. Πολλές φορές έχουμε το εμπόρευμα αλλά δεν έχουμε το μαγαζί που θα το πουλήσει. Και θα πρέπει βέβαια αυτές τις ταινίες να προβάλλονται επί περισσότερο χρόνο. Άρα υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας στις αίθουσες από πλευρά των ευρωπαϊκών ταινιών που είναι μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος γιατί έχουμε αυτό το τρομερό δίκτυο στην Ευρώπη το οποίο όμως δεν έχει ε, προπολογισμό αρκετό στη διάθεσή του οπότε θα πρέπει πολλά να φροντίσουμε όσον αφορά την ε, διανομή των ταινιών. Αυτά είχα να σας ε, προτείνω και ευχαριστώ να απαντήσω αν τυχόν έχετε κάποιες ε, ερωτήσεις. Ο Βίμ δεν ήθελε να μιλήσει τώρα στις λεπτομέρειες της διανομής, εγώ θα προσπαθήσω να σας πω τις προτάσεις μου. Είναι πρακτικό χαρακτήρα. Λεπτομερείς, συγκεκριμένες, αλλά σημαντικές. Έχουμε περισσότερα έργα ευρωπαϊκά στις οθόνες. έχουμε περισσότερους κινηματογράφους που να δείχνουν ευρωπαϊκά έργα. Να υπάρξουν περισσότεροι πόροι για να βελτιωθούν οι υπάρχουσες αίθουσες, να ανακαινιστούν. Περισσότερες οθόνες, καινούργιες οθόνες. Σε πολλές χώρες αυτό δεν γίνεται εάν δεν υπάρξουν κονδύλια ευρωπαϊκά. Επίσης να δούμε εάν μπορέσουμε να έχουμε και επιπλέον μέτρα για να γίνει το ευρωπαϊκό σινεμά πιο ελκυστικό. Να έχουμε κίνητρα για τους κινηματογράφους για να δείχνουν ευρωπαϊκές ταινίες. Κυρίως τις ταινίες του Μίντια. Οπότε θα πρέπει να αυξηθεί το σχετικό ευρωπαϊκό κονδύλιο. Και έτσι να έχουμε κάποιο ποσό ικανοποιητικό. Τώρα κάτι γίνεται αλλά είναι πιο πολύ για το Θεαθήνα, δεν είναι τόσο πολλά χρήματα. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει και με τους πόρους του Μίδια γιατί έτσι βοηθούνται οι διανομής. Έτσι πείθονται οι αίθουσε να προβάλλουν κάποιες ταινίε περισσότερο χρόνο. Γιατί οι ταινίες καλλιτεχνικής ποιότητας ε, δεν μπορούν να συναγωνιστούν ε, στα αμερικάνικα blockbusters και χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να τα μάθει ο κόσμος. Ξέρετε τι είχε πει ο διάσημος Βρετανός δημιουργός Κεντ Λόουις. Είχε έρθει σε ένα πάνελ στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου και ξέρετε τι είπε. Κάτι με το οποίο συμφωνώ. Ότι ό,τι κάνουμε με την όπερα και με το θέατρο, το κάνουμε και με το σινεμά. Θα πρέπει οι δήμοι και οι κοινότητες να αναλάβουν τα ενία θα πρέπει να ασχοληθούν κάποιοι που αγαπούν τον κινηματογράφο και όχι κάποιοι που ασχολούνται με το fast food γιατί πολλές φορές τη διαχείριση των κινηματογράφων την έχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Άρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα δοκιμαστικό πιλωτικό πρόγραμμα. Και έτσι να έχουμε κέντρα κινηματογράφου ελκυστικά κινηματογράφου ελκυστικούς με πολλές οθόνες. Ένα πρόγραμμα που να καλύψει στην αρχή ε, κάποιους κινηματογράφους της μεγαλύτερης πόλη τη Ευρώπης, κυρίως εκεί που το μερίδιο των είναι που δείχνεται δεν είναι πολύ μεγάλο. Τι άλλο, άλλο. Να σας πω τι έχει πει ο Πιότρο Μπόρις είναι από το Βρόσλαφ, είναι ευρωβουλευτής και πριν έρθει εδώ να γίνει ευρωβουλευτής ήταν περιφερειάρχης κάπου στην Πολωνία και είχε αρμοδιότητες πολιτιστικές και χάρη στο έργο που επετέλεσε στο ε, υπό εκεί που πριν δεν είχαμε κανένα κινηματογράφο ποιότητος χάρη σε αυτόν πήρε έναν κινηματογράφο 700 θέσεων και το ανακαίνισε, το έκανε multiplex με mediatek, με βιντεοθήκη, με καφέ, με πολλές οθόνες και εκεί προβάλλονται ευρωπαϊκές ταινίες. Η επένδυση ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ, το 30% καλύφθηκε από τα διευθυντικά ταμεία, η διαχείριση έγινε από την κυβέρνηση και την τοπική, ε, τοπικές αρχές και τα υπόλοιπα είναι κονδύλια του Βρότσλοφ. Από αυτούς που είναι ιδιοκτήτες του σινεμά αυτού του κέντρου. Να, επομένως, να παράδειγμα προς μίμηση, πώς μπορεί να συνδυαστεί η τοπική πρωτοβουλία με την ευρωπαϊκή βοήθεια. Επομένως, θα πρέπει και ο να χρησιμοποιηθεί για να εκπαιδεύσει το κοινό και θα πρέπει να έχουμε ένα οπλοστάσιο με ταινίε, ευρωπαϊκές, μίνι φεστιβάλ, ε, συνεκριτικές και όλα αυτά θα πρέπει να σε στενή συνεργασία με τους διανομής. Μην ξεχνάμε ότι οι διανομής είναι πάρα πολύ σημαντικοί για όλη αυτή την υπόθεση, γιατί αυτοί εξασφαλίζουν την διάδοση των ευρωπαϊκών ταινιών. Πολλές φορές είναι συμπαραγωγή. Διαχειρίζονται τις αίθουσε και οργανώνουν φεστιβάλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα βοήθησε την ψηφιοποίηση. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Όλα αυτά που σας λέω εδώ δεν αφορούν όλα τα θέματα διανομής. Απλά εισαγωγικά σας τα λέω. Γιατί θα πρέπει να γίνει ένα σοβαρό προβληματισμό και να αναζητήσουμε τον τρόπο ο Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο να μπορέσει να προσαρμοστεί στου μοντέρνου καιρού. Λοιπόν, μα δώσατε διάφορα θέματα που θα μπορούσαμε του επόμενου μήνε ίσω να λάβουμε υπόψη για τι συζητήσει μα για να πετύχουμε του στόχου που αναφέρατε και οι τρει. Πριν περάσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα ακόμα να δώσω το λόγο στο φίλο μας από την Ιταλία, στον Τέοντιο Κοσέτη, γενικό στους ε, Venice Days. Να πω δύο λόγια ακόμα. Οι μέρες αυτές της Βενετίας, Venice Days, είναι κάτι θαυμάσιο μέσα στα πλαίσια της Μόστρα τη Βενέτσια. Και πρόκειται για τις μέρες των δημιουργών, που μας βοηθήσαν πάρα πολύ φέτος γιατί στις Κάνες είχαμε την ιδέα να έχουμε ένα κοινό σχέδιο, το, το βραβείο Λουξ και τις ημερίδες αυτές ε, στην Βενετία. Καλήσαμε 27 ε, νέους από κάθε κράτος χώρας ένα. Τους καλέσαμε, τους πληρώσαμε ταξίδι και τη διαμονή τους. Και αυτό ήταν το πρώτο σχέδιο ε, 27 χρόνια από τον κινηματογράφο και είδανε κάποιες ταινίε, συζητούσαν τις ταινίε αυτές από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέσω διαδικτύου συζητήσαν για τις ταινίε αυτές θαυμάσια συνεργασία. η κυρία Κώστα Οσκουρία και οι υποφαινόμενοι ήμασταν εκεί την Παρασκευή, την πρώτη τελευταία ε, μέρα, δηλαδή στο λεγόμενο αυτό ε, τμηματικό κινηματογράφο των 27 και ο Βιμβέντερς που είπε αν τους είχα εγώ αυτούς τότε θα έκανα θαύματα. Δεν μπορεί κανένας πραγματικά να εκτιμήσει τι σημαίνει. Γιατί αυτοί οι νέοι μεταδίδουν αυτή την ιδέα σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η, μια ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, ημερών αυτών στη Βενετία μαζί με το βραβείο Λούξο που προχωρήσε κοράμε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολύ την Ευρώπη, ούτε καν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε και το Κοινοβούλιο δεν κάνει και τίποτα. Αλλά τώρα θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Τζόρια Κοσέτη που μπορέσαμε να έχουμε τους ανθρώπους αυτούς εκεί, τους νέους εκεί. Έχετε το λόγο, Τζόρια. Yes, Mr. President. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Και υπόσχομαι να τηρήσω το χρονικό όριο των 10 λεπτών. Και φυσικά θα μιλήσω στα Ιταλικά. Γιατί είμαστε υπερήφανοι εμεί οι Ιταλοί, ιδίω σε αυτή την εποχή. Ακου, ακούγοντας ε, ε τα, όσο, τα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί, ε, επιβεβαιώθηκε η άποψή μου ότι ίσως ο χειρότερος εχθρό της Ευρώπης και του πολιτισμού της Ευρώπης είναι ίσω η Ευρώπη. Έχει δίκιο ο Βιμβέντερ που λέει όταν γυρνάει τον κόσμο, ότι αισθάνεται κανείς υπερήφανος που ε, αποτελεί μέρος και συμμετέχει στην ε, ευρωπαϊκή κουλτούρα. Έχει δίκιο ο που λέει ότι ο πολιτισμός μας και η Ευρώπη ολόκληρη στην πραγματικότητα από όλο τον κόσμο θεωρείται κάτι το σημαντικό, κάτι που προσφέρει αξία. Έχουν δίκιο αυτοί που μίλησαν σήμερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κινηματογράφος. Και όταν λέω ότι είμαστε οι εχθροί του κινηματογράφου μας και του πολιτισμού μας, ε, σκέφτομαι τις εθνικές κυβερνήσεις που στην πραγματικότητα δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν μεταξύ τους ούτω ώστε ο κινηματογράφος να μπει μέσα στο πρόγραμμα των σχολείων. Ούτε είναι ικανές να συμφωνήσουν μέσα στα κράτη ε, στο να γίνει ο κινηματογράφος η οικαστική μνήμη της ιστορίας μας γιατί κάθε ε, εθνικός την, αφηγείται την ιστορία του κράτους αυτού, την ιστορία της Ευρώπης. Ένα υπέροχο εργαλείο για να καταλάβουμε το παρελθόν μας. Και δεν είμαστε ικανοί να το αξιοποιήσουμε. Δεν είμαστε ικανοί, ούτε εσείς ίσως, κύριε Ευρωβουλευτές, δεν είστε ικανοί να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι η έννοια της Ευρώπης η πίστη της για... στην Ευρώπη ανάμεσα στους πολίτες. Όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως, αλλά για την Ευρώπη την ίδια. Ναι, εκεί ζούμε. Ε, η κυρία Ντόρις Μπακ ε, είχε την ε, ε, ευγένεια ε, να μιλήσει τόσο θετικά για αυτή την πρωτοβουλία του, που είχε το τίτλο 27 Times Cinema που υλοποιήθηκε στη Βενετία. Αυτά όμως τα 27 παιδιά που ήρθαν και που ήταν μόνο ένα σπόρος, μια ένδειξη για όλα αυτά που μπορούν να γίνουν. Ρωτήστε, τον Νίκολα Σό και τον Τόμα Σμόλτερ που βρίσκονται εδώ σήμερα παρόντες και τους ευχαριστώ. Ρωτήστε τους, θα σα πούνε ότι διασκέδασαν. Με μεγάλη χαρά ανακάλυψαν τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Αισθάνθηκαν κατεξοχήν κομμάτι μιας ε- Ευρώπης, χωρίς ανάγκη καμιά ρητορίας. Ήταν προφανή η Ευρώπη. Εγώ λοιπόν θα περιοριστώ ε, στην ε, παρουσίαση μου αυτή να μιλήσω για τα φεστιβάλ. Είμαι κατασκευαστής φεστιβάλ. Πριν έρθω εδώ α, αντάλλαξα ε, απόψεις με τον ε, ε Τσάγκο Ματζόρε με τον οποίο συμμετέχουμε, με τον οποίο συμμεριζόμαστε την ίδια ιδέα και την ίδια επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι στην Ευρώπη και είπαμε ότι τα φεστιβάλ είναι ένα άλλο κομμάτι αυτής της συζήτησης που άνοιξε σήμερα με τόσο σημαντικό και συγκεκριμένο τρόπο και σας παρακαλώ να μείνετε σε αυτό το συγκεκριμένο, το χειροπιαστό επίπεδο. Τα φεστιβάλ είναι ένας τρόπος κατάρτισης του κοινού. Αυτή τη στιγμή χάνουμε δυστυχώς το πρώτο μέσο που υπάρχει που είναι το σχολείο. Για μένα είναι σημαντικό να μην χάσουμε και το δεύτερο μέσο που είναι τα φεστιβάλ. Υπάρχει το δίκτυο Euro ένα δίκτυο ε, κινηματογραφικών αιθουσών που είναι ε, ένα εξαιρετικό δείγμα ζωτικότητας που, για το οποίο μας μίλησε και ο Ρόμαν Γκούτεκ. Ε, τα φεστιβάλ πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Η γενιά του Βιν η δικιά μου, μεγάλωσε μέσα στα φεστιβάλ που ήταν για μας τόποι ανακάλυψης ε, γνώσης συνέστησης όπως ήταν και ο κινηματογράφος όπως ήταν και οι ταινιοθήκες ε, στην εποχή μας. Σήμερα τα φεστιβάλ κινδυνεύουν να γίνουν γκλάμουρ, ε, κόκκινο χαλί, ένα είδος τηλεοπτικού τύπου μια πλατφόρμα ε, του κινηματογράφου. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού του πράγματος, αλλά πιστεύω ότι είναι καθήκον αυτών που φτιάχνουν τα φεστιβάλ ε, να μην ξεχνάνε ότι πρέπει το φεστιβάλ να είναι τόπος ανακάλυψης και γνώσης. Από το Αμπου Τάμπι έως τη Σαγκάη, από το Μπένος Άιρες μέχρι στο Ουαγκαντουγκού, η απάντηση είναι παντού η ίδια. Μας ενδιαφέρει ο ποιοτικό κινηματογράφος. Και ο ποιοτικό κινηματογράφος, κυρίες και κύριοι, πολύ συχνά σε ολόκληρο τον κόσμο είναι συνώνυμο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος των συμπαραγωγών, του ανοιχτού πνεύματος, που δεν είναι ο βαρετός κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος του Wim Wenders δεν είναι βαρετός κινηματογράφος. Τον ξέρει όλος ο κόσμος. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος πρέπει να είναι υπερήφανος και πρέπει να προ προωθηθεί σαν ένα στόχος προς επίτευξη. Κοιτάζω και το ρολόι μου και σας λέω απλώς ότι το να καταρτιστεί το κοινό πρέπει να είναι και είναι το συγκεκριμένο καθήκον μας. Να καταρτήσουμε το κοινό. Τι σημαίνει να του δώσουμε τις ευκαιρίες και την περιέργεια να κάνει κάτι. Η ε, εμπειρία του 27 Times Cinema έδειξε ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει 27 άτομα μέσα σε ένα τεράστιο φεστιβάλ όπως είναι η της Βενετίας. Τίποτα. Είναι όμως ο σπόρος, ο ιδεολογικός και πολιτικός, ε, μια συγκεκριμένη ένδειξη για το τι μπορεί να γίνει. Και πέρασαν αυτές τις μέρες όχι μόνο διασκεδάζοντας, αλλά και αποκτώντας την αγάπη για το φεστιβάλ σαν ε, τόπο γνώσης και ανακάλυψης. Ε, να τελειώσω λέγοντας το εξής. Είπαμε και ρωτήσαμε, αναρωτηθήκαμε μεταξύ μας, τι μπορούμε να πούμε εμείς, οι άνθρωποι του κινηματογράφου, στους ανθρώπους της πολιτικής. Λέω λοιπόν το εξής. Να ε, διασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα τους θησαυρού που έχουμε. Το πρόγραμμα Media είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρό. Χωρίς το πρόγραμμα Media, πολλά φιλμ σημαντικά, όχι μόνο βραβευμένα, αλλά και αυτά που έχουν χειροκροτηθεί από το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα υπήρχαν σήμερα. Χωρίς τις πρωτοβολίες του Media και το διεθνές του άνοιγμα, δεν θα υπήρχε ακριβώς μια δουλειά όπως το Europa, το Ευρώπα Σινεμά, ε, όλα αυτά τα μέσα διανομής, κυκλοφορίας και γνώσης που αυτή τη στιγμή εμείς οι επαγγελματίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σίγουρα μπορούν να γίνουν καλύτερα πράγματα και πρέπει να κάνουμε καλύτερα και πάντα πρέπει να ζητάμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά να είστε υπερήφανοι για αυτό που έχετε και να το υποστηρίζετε. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τον πολιτισμό στο επίκεντρο των προσπάθειών της λόγω και των οικονομικών δυσκολιών. Όμως υπάρχουν ε, προσπάθειες σε όλη την Ευρώπη που μας δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Να πω δύο λόγια ακόμα για το βραβείο Λουξ. Τα βραβεία ο Βιμ Βέντερς αναφέρθηκε στην Ακαδημία, που είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός στην Ευρώπη. Το βραβείο Λούξ είναι κάτι το πολύ πιο πρόσφατο. Βραβείο δεν σημαίνει χρήματα. Δεν σημαίνει αυτόματα αναγκαστικά ποιότητα. Σκεφτούμε τα Όσκαρ. Αλλά το βραβείο Λούξ, που είναι το δικό σας βραβείο, πριν ακόμα δημιουργηθεί, βράβευσε τον Φάτι Ακίν που ήταν ακόμα πολύ νέος. Βράβευσε το Welcome, ένα από τα ευρωπαϊκά έργα που γύρισαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ε, φιλμ ολόκληρη την Ευρώπη. Τα, από τα τρία πρώτα φιλμ που βραβεύσατε, τα δύο ήταν υποψήφια για Όσκαρ ξένης ταινίας. Δεν σημαίνει ίσως τα πάντα αυτό που σας λέω, όλα σημαίνει κάτι. Σημαίνει κάτι που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Λοιπόν, εμείς αυτό με το 15η ημέρο, με τις ημέρες του, των δημιουργών στη Βενετία, ε, θέλουμε ε, ακριβώς μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες μας να θέσουμε σε κυκλοφορία τα βραβεία Lux. Με μία προϋπόθεση. Το καθήκον μας σαν φεστιβάλ είναι να απευθυνθούμε σε ένα κοινό νεανικό, να μιλήσουμε στους νέους, να μην κλειστούμε ε, μεταξύ των δημιουργών, να μην πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε η ελίτ. Ο Ρόμαν Γκούτεκ μας ε, υπενθύμησε ότι το θέατρο και η όπερα ήταν ε, τελείως λαϊκά ε, μέσα για έναν ολόκληρο αιώνα το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον κινηματογράφο. Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία, ανοιχτή σε όλους. Κοιτάξτε, ο κόσμος έρχεται στον κινηματογράφο. Οι εθνικοί κινηματογράφοι γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς και σημαντικοί στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί είχαν το θάρρος να απευθυνθούν στο κοινό τους. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος πρέπει να κάνει το ίδιο. Πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του. Εμείς ευχαρίστως θα ε, κάνουμε το καθήκον μας από την πλευρά ε, των φεστιβάλ ε, πιστεύουμε ότι πρέπει τα φεστιβάλ να έχουν μια υποστήριξη όχι μόνο οικονομική αλλά και θεσμική, κανονιστική από το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν χρειαζόμαστε τόσο χρήματα όσο το κύρος της Ευρώπης που πρέπει να σταθεί στο πλευρό αυτών που ασχολούνται με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ε, του κοινού. Ελπίζω να σας είπα κάτι συγκεκριμένο. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ε, δεν ε, ε, αρκεί ένα πρωινό όπως το σημερινό. Αλλά αν θέλουμε να παίρνουμε σπόρους σαν αυτό του 27 Times Cinema της Βενετίας, πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε με τρόπο συγκεκριμένο και έξυπνο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι. Γιατί και η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να μιλήσουν και ελπίζω να μην μακρηγορήσουν. Σίγουρα κατέγραψαν όλα όσα ελέγχθησαν. που κατά μεγάλο ποσοστό απευθύνεται προ τα κράτη-μέλη και προ την Κομισιόν επίση. Η Μαρία Πατιακούτση έχει το λόγο. Πρόεδρε, Έχοντα ακούσει του ομιλητέ έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος brainstorming, συλλογής ιδεών. Τόσο πολλές είναι οι ιδέες που ακούσαμε εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε κάποια συγκεκριμένα λίγα σημεία μόνο. Ε, όλοι συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση για τον κινηματογράφο είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα, αλλά και τους μελλοντικούς καταναλωτές του κινηματογράφου. Και αυτούς που διδάσκουν το προσωπικό των κέντρων ε, εκπαίδευση. Όλοι αυτοί να είναι εκπαιδευμένοι στα οπτικοακουστικά, τα καινούργια, γιατί όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι τόσο να χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο για να διδάξουν ε, το, το, την ιστορία, οποιοδήποτε άλλο μάθημα και γι' αυτό βασικά θέλω να, να δούμε τι θα κάνουμε με τους ανήλικους, τους έφηβους, τους μικρούς και η ερώτησή μου είναι η εξής όλοι αυτοί μικροί έφηβοι και αυτοί χρησιμοποιούν κάποια καινούργια σχήματα, καινούργια μέσα, καινούργια ε, συσκευές ε, για, τις, ε, για, για κινηματογράφο, για σπορ, για οτιδήποτε θα πρέπει το περιεχόμενο πολλές φορές ε, είναι πολύ βίο το περιεχόμενο σου και να θέλουμε να μην είναι. Οπότε τι θα κάνουμε. Οι διάσημοι σκηνοθέτε οι συγγραφείς, αυτοί που δημιουργούν τον πολιτισμό στην Ευρώπη, πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν ούτως ώστε το περιεχόμενο αυτών των gadget που χρησιμοποιούν οι μικροί να είναι κάτι το ποιοτικό κάτι το οποίο να βοηθάει και την εκπαίδευση και ταυτόχρονα να δημιουργούνται έτσι οι μέλλοντες συντελεστές του κινηματογράφου και βεβαίως έτσι να μπορούμε να δημιουργούμε πολίτες να δημιουργούνται κάποιο συνέργεια μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ Μαρία. Ο επόμενος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις σκέψεις σας όσον αφορά τον πολιτισμό στην Ευρώπη και επίσης για τον κινηματογράφο που μας μιλήσατε για την παιδεία, την καλλιτεχνική παιδεία των νέων και πώς μέσω από εικόνες θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό που θέλουμε. Να, τι θα πρέπει να έχει προτεραιότητα στις ιδέες μας όπου θα ασχοληθούμε με τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εδώ και λίγες εβδομάδες είχαμε κοινωνιολόγους που ήρθαν και μας εξήγησαν και κάποιες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες η μεγάλες αλλαγέ συμβαίνουν όχι κάθε 20 χρόνια όπω κάποτε, αλλά κάθε 7 χρόνια. Αλλάζουν οι γενιέ. Ο κύριο Καβαντά, ο ούγρος ε, συνάδελφο μας είπαν για τους κινδύνους που εγκυμονούνται αν δεν έχουμε κάποια αισθητική υπέρ του κινηματογράφου. Αναφέρθηκαν και κάποια παραδείγματα. Μιλήσαμε για κάποια φεστιβάλ με 100.000 ε, επισκέπτες σε 7 μήνες αρχίζει η Πολωνική Προεδρία. Εμείς θα την προσοχή μας στην παιδεία, στον πολιτισμό και στον κινηματογράφο. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτών των πρωτοβουλειών του Βιμ Βέντερς και έτσι να ελκύσουμε τον πρόεδρο Μπαρόσο και την προσοχή του. Να βοηθήσουμε τους νέους να προσπαθήσουμε να ψηφιοποιήσουμε τον κινηματογράφο και έτσι μέσω του ψηφιακού κινηματογράφου οι διανομής να μπορέσουν να μοιράσουν παντού τα έργα τους και να είναι πιο ελκυστικός ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Ευχαριστώ. Κύριε Μπίσκη, έχετε το λόγο. Μια που ηγείστε και κάποιες Ροφικής ακαδημίες στη χώρα σας. Μας τα είπε ο κύριος Βέντερς, μας μίλησε για το ρόλο της γλώσσας. Τι γίνεται με τη μετάφραση, έχουν ληφθεί κάποια ενθαρρυντικά μέτρα. Γιατί πολλοί φορές λείπουν τα χρήματα για κάτι τέτοιο. θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ίσω τεχνολογία. Δεν λέω να δαπανίσουμε πάρα πολλά, απλώς να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να βοηθήσει. Κάτι άλλο τώρα, κάτι το οποίο ήδη κάποιος το έδειξε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε τους δάσκαλους, τους καθηγητές στη Γερμανία. να έρθει ο κόσμος στο Ίδρυμά μας, το Μπάμπλεσμπεργκ, και να δει τις στολές, τα κουστούμια. Όλοι όσοι έρχονται εκεί πολλά μαθαίνουν, αλλά να μπορέσουμε να στοχοθετήσουμε κάποιους όπως τους ε, καθηγητές για να περάσουν αυτά τα μηνύματα. Νομίζω ότι αυτό κάτι μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και ακούω όλα αυτά τα θετικά μηνύματα από τους ομιλητές μας και ιδιαίτερα του κυρίου Βέντερς που έχει ε, συμβάλει σε τεράστιο βαθμό στην ε, υπόθεση αυτή με τις ταινίε του. Το ευρωπαϊκό όνειρο, κάτι παρόμοιο με το αμερικάνικο όνειρο, αναφέρθηκε. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω όμως, και είναι μια ερώτηση, είναι το εξής. Το αμερικάνικο όνειρο ήταν εύκολο να δημιουργηθεί, ευκολότερο, γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση και μια γλώσσα. Εμείς έχουμε 27 κράτη-μέλη, σχεδόν τον ίδιο αριθμό γλωσσών, και αναρωτιέμαι, υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερο υποτιδλισμό των έργων ή για voice over. Ε, γιατί έτσι ε, μπορεί να ακουστεί και ε, η προφορά των ανθρώπων που απεικονίζονται. Είναι ένα δίλημα αυτό. Και η σχετική χρηματοδότηση. Θα ε, κάτι άλλο. Θα έπρεπε να σκέφτεται κανεί το ευρωπαϊκό όνειρο ή την ευρωπαϊκή κραυγή, European Dream or European Scream. Ε, κάτι άλλο για τα φεστιβάλ. Όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, και βεβαίω τα δεχόμαστε. Ε, ε, ίσως θα μπορούσατε να επεκταθείτε περισσότερο πάνω στο θέμα του βραβείου Lux. πώς θα μπορούσε να γίνει πιο χρήσιμο και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το βραβείο Λούξ ε, ή το μεταγλωτισμό, το voice ε, σήμερα έχουμε εδώ μια ομάδα φοιτητών. Ε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για αυτούς να ακούν αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια από ανθρώπους της ε, δικιάς σας ποιότητας, του δικού σας διαμετρήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλωσορίζουμε τους Ιρλανδούς φοιτητές, λέει η Πρόεδρος, και όλους τους άλλους. Ο κύριος Μπάργκο είναι ο τελευταίος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι υπέροχο να συμμετέχει κανείς σε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την εκδήλωση. Καλύπτει ένα τεράστιο κενό Αναρωτιέμαι ε, αν μια συζήτηση τέτοιου μεγέθους, τέτοιων διαστάσεων είχε οργανωθεί ε, στο πρόσφατο παρελθόν του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ανάμεσα στους, ε, στο πολωνικό και στον ουγγρικό λαό παραδοσιακά μια φιλία και γι' αυτό αισθάνομαι πιο κοντά στον κύριο Ρόμαν Γκούτετς δεν θέλω να στρουθώ καμιλίζω, θέλω να ε, υιοθετώ πάντοτε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτό που βλέπουμε ε, σήμερα είναι ότι η τέχνη είναι χαμένη πάντοτε σε σχέση ε, με, την επιχειρηματικότητα. Άρα δεν θα πρέπει να λυπόμαστε τους ε, ανεξάρτητους δημιουργούς. Υπάρχει μια ουγγρική παροιμία που λέει ανάμεσα στον ε, τρελό και στη μεγαλοφία ε, υπάρχει στην τέχνη μόνο μία διαφορά και αυτή είναι η επιτυχία. Αν δούμε ε, το, το θέμα της, από την οπτική γωνία της επιτυχίας, το Star Wars και τα λοιπά, Πρόσφατα είχα μια συζήτηση όπου πληροφορήθηκα ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι ε, ζωντανός, ε, είναι καλύτερα ε, από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή είναι η κληρονομιά μας και την έχουμε αναγεννήσει. Πρέπει να σταθούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και γι' αυτό αναφέρομαι στις προηγούμενες ερωτήσεις που έγιναν ε, σχετικά με τη χρηματοδότηση και το μάρκετινγκ. Αλλά λάβουμε υπόψη μας τον προϋπολογισμό των ε, ε, παραγωγών του Χόλιγουτ είναι μεγαλύτερη από το εθνικό εισόδημα κάποιων μικρών δημοκρατιών. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες, ε, ε, κάποιες πρόσθετες αξίες ε, που δεν θα πρέπει να παραμελούνται μέσω του ισοποδοτικού μάρκετινγκ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία γραπτή, συγκεκριμένη στρατηγική και χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω στους κυρίους αυτούς τη δυνατότητα να απαντήσουν στι ερωτήσει ή στι αντιδράσει που ακούστηκαν. Θέλετε κάτι να πείτε? Όχι? Κύριε Κοζέτη, θέλετε κάτι να προσθέσετε ή απλώς σας ικανοποιήσουν αυτά που ακούσατε. Νομίζω ότι είπατε τα πάντα πάρα πολύ καλά. Είναι μια στιγμή κοινή σκέψη θεωρώ, δεν το τόνισα ίσω ότι η σημασία τη εφαρμογή από το Κοινοβούλιο του σχεδίου 27 Times Cinema 27 φορέ κινηματογράφο, είναι ουσιαστικό γιατί αυτό καταδεικνύει τι μπορεί να γίνει και δίνει συγκεκριμένα μηνύματα στρατηγικές σχεδίων που μπορούν πραγματικά να εφαρμοζούν και να αλλάξουν την ε, στάση της νεολαίας. Θα πρέπει την νεολαία να μην την καταστρέψουμε, να της μιλήσουμε κατάματα. Μετά τις σημερινές συζητήσεις, θα ήθελα να τονίσω σημασία του φεστιβάλ. Όσο πάει υπάρχουν περισσότερα φεστιβάλ. Εγώ περνάω τις διακοπές μου στην Ορμανδία και υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός μικρών φεστιβάλ, ακόμη και ένα μικρό φεστιβάλ ευρωπαϊκού κινηματογράφου, όπου υπάρχουν όσο πάει και περισσότεροι νέοι θεατές και μου φαίνεται είναι θαυμάσιο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω στο ρόλο αυτό των φεστιβάλ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Jeszcze sekundkę, żeby odpowiedzieć na te pytania dotyczące tłumaczeń. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας για τις ε, μεταφράσεις, τους μεταγνωματισμούς των ε, ταινιών. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο χρηματοδότηση, γιατί στο πρόγραμμα Μέντια που υποστηρίζει τη διανομή υπάρχουν χρήματα για, την, ε, για το μεταγλωτισμό ή τους υπότιτλους. Και στα φεστιβάλ επίση υπάρχει δυνατότητα εκ των εσόδων να χρηματοδοτηθεί αυτό. Για τα φεστιβάλ έχω να πω ότι πολλές φορές τα φεστιβάλ είναι η μόνη δυνατότητα ε, να δει κανένας ε, τους ταινίες αυτές σε μία ε, οθόνη κινηματογράφου. Γιατί πολλές από αυτές τις ταινίες δεν τη βλέπει κανένα σε, σε οθόνη κινηματογραφική. Να επανέλθω σε αυτό το φεστιβάλ του Αμερικανικού κινηματογράφου που οργάνωσα και που έληξε πριν από μερικέ μέρες. Περιέργως όταν έρχονται για να δουν μια αμερικανική ταινία είναι πολύ πιο εύκολο μέσω αυτού να ενδιαφερθούν για τον κινηματογράφο και ε, μετά με την παράδοση των ετών ενδιαφέρονται και για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Έχω μια πρόταση κύριε Μποτέκ, Κάντε ένα φεστιβάλ για τι ευρωπαϊκές εταιρείε που δεν έχουν ειδωθεί, όχι μόνο για ανεξάρτητε αμερικανικές, αλλά για εξάρτητες ε, ταινίε ευρωπαϊκές που δεν έχουν ακροματικότητα. Εντάξει, καλή ιδέα θα ήταν αυτό. Ε, ναι, να σας ε, οργανώσουμε ένα τέτοιο φεστιβάλ στο Φάλσοφ τον Ιούλιο δείχνουμε 70% ευρωπαϊκών ταινιών σύμφωνα με τις απαιτήσει του προγραμμάτος Media. Και φέτος είχαμε 120.000 θεατές. Αυτή είναι η απάντησή μου. Πολύ ωραία. Ο κύριος Φέντας και εγώ αναφερόμενο στο θέμα των γλωσσών. Η ψηφιοποίηση των κινητών οθονών καθιστά πολύ πιο εύκολη τη χρήση γλωσσών. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχει κανένα μόνο μία γλώσσα με υπότιτλους. Αλλά ένα μια ψηφιακή ταινία μπορεί να έχει πολλές γλώσσες που να ανοίγουν και να κλείνουν με ένα κουμπί και μόνο. Ο μετακροτισμός χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες. Στην Ιταλία οι περισσότερες ταινίες είναι μετακροτημένες. Στη Γαλλία μειώνεται. Πριν από λίγο καιρό είχαν 50% περίπου των ταινιών και τα 50% είχαν υπότιτλους, σήμερα ακόμα και ε, σε ε, χώρες στην, ε, στην περιφέρεια χρησιμοποιούν πραγματικά τους υποτίτλους. Είναι γι' αυτό ένας τρόπος παιδείας. Εμείς είμαστε υπέρ των υποτίτλων. Και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών ταινιών. Δύο λόγια για την Ακαδημία μας, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Εμείς υπάρχουμε μόνο και με μόνο στόχο να προωθούμε, να γιορτάζουμε τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Εμείς ταξιδεύουμε κάθε δύο χρόνια σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε στην Ιταλία. Ε, θα δώσουμε τα βραβεία που θα μπορεί να δει κανένα στην ε, τελετή της βράδευση σε 46 χώρες στην Ευρώπη και μέχρι την Ιταλία. Αυτό χρηματοδοτείται σε μεγάλο ποσοστό από το, την πόλη του Βερολίνου, τα βραβεία από διάφορους πόρους και έτσι βοήθησε η Ακαδημία αυτή να προωθήσει τον ε, Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Αν μπορώ να σας δω ε, εκεί, ε, θα χαρώ πολύ. Αν μπορείτε όλοι να έρθετε στην Ιταλία, θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ να σας δω. Να σας ευχαριστώ. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ το Vivenders. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο για σύντομες παρεμβάσεις σε κάποιον εκπρόσωπο της Βελικής Προεδρίας, σε έναν από τους δύο, είστε δύο, αλλά παρα, παρακαλώ ένας να μιλήσει μόνο. Ποιος? Ο κ. Μπλονσάχ. Θα προωτούσε η κυρία να μιλήσει, αλλά νομίζω ο κύριος Μπλανσάρ είναι για, την, για τον πολιτισμό και η κυρία είναι για την εκπαίδευση. Παρακαλώ, πέντε λεπτά. Euh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που μας καλέσατε σε αυτή την ακρόαση που ήταν πραγματικά συναρπαστική και ε, πιο προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα που είχα την ευκαιρία να συναντήσω ε, τον σκηνοθέτη της ταινίας αυτής ε, «Τα φτερά του έρωτα» στα ελληνικά, στον ουρανό του Βερολίνου που με συγκλώνησε πραγματικά κατά τη δεκαετία του 80. Ε, θα μιλήσω, θα δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου τη Ζάννα Μπραφό ε, να σας μιλήσει για την Προεδρία και για τις προθέσεις Προεδρίας ε, με βάση μια άτυπη σύσκεψη των Υπουργών που έγινε εδώ τον Οκτώβριο και εγώ θα σας μιλήσω για τα πιο επίσημα προγράμματα της Προεδρίας και όσα πρόκειται να συζητηθούν στο Συμβούλιο τον Νοέμβριο. Λυπούμε, λοιπόν, δεν μπορείτε να δώσετε εσεί το λόγο σε κάποιον άλλο. Εγώ σε έδωσα σε εσά το λόγο. Έτσι. η συνάδελφό σα και εσείς θα μιλήσετε μετά. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Okay, no, euh, euh, très brièvement, donc, euh, Ωραία, πολύ σύντομα τότε. Μία από τις ε, πολιτικές προϊόντες της Προεδρίας μας ήταν η δημόσια υποστήριξη του κινηματογράφου. Τον Ιούλιο οργανώσαμε ένα συμπόσιο ε, ε, και ακολούθησε μια άτυπη σύνοδο των Υπουργών τον Οκτώβριο και ο σκοπός ήταν ακριβώς να ε, επιβεβαιώσουμε την σημασία της δημόσιας υποστήριξης για τον κινηματογράφο. Γιατί χωρίς δημόσια υποστήριξη νομίζουμε ότι δεν θα, υπάρξει, δεν θα υπάρχει ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την ε, αναθεώρηση της ε, ανακοίνωσης για τον κινηματογράφο που ρυθμίζει διάφορα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιμένοντας ε, όλος ιδιαιτέρως στο θέμα ότι η δημόσια στήριξη δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την κινηματογραφική παραγωγή αλλά όλα τα στάδια της αλυσίδας. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική κινηματογράφου παρά μόνο να δούμε τον κινηματογράφο στο σύνολό του. Όσον αφορά το τι θα γίνει στο Συμβούλιο εκπαίδευσης ε, νεολαίας και πολιτισμού τον Νοέμβριο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε υποβάλει δύο σχέδια συμπερασμάτων ε, που είναι αρκετά ευθυγραμμισμένα με, τη, με το νόημα της συζήτησης που έγινε σήμερα. Ε, το θέμα ε, της ψηφιακής εποχής είναι το ένα θέμα σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και πώς μπορεί να διατηρηθεί ε, η κληρονομιά αλλά και να υπάρχει πρόσβαση στην κτηματογραφική κληρονομιά ε, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και πόσο σπουδαίο είναι για τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για την κτηματογραφική κληρονομιά ε, η γνώση της πολιτικής κληρονομιάς είναι κάτι το θεμελιώδες για την κατανόηση του κινηματογράφου για την κινηματογραφική παιδεία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ε, βλέπουμε το σημερινό κινηματογράφο χωρίς να έχουμε γνώση του, των διαφόρων καλλιτεχνικών ρευμάτων, της Νουβέλ Vague, του ε, νεορελισμού, της Ιταλίας κλπ. Μετά, η δεύτερη ανακοίνωση το δεύτερο ε, συμπέρασμα, σχέδιο συμπεράσματο, αφορά μια ανακοίνωση τη ε, Κομισιόν ακριβώ για την ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αιθουσών. Υπάρχει σχετικά λοιπόν η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης της Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι η Κομισιόν θα μας μιλήσει γι' αυτό στη συνέχεια. Ε, τονίζεται ε, το γεγονό ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή γίνεται κάτι το επίγον και είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν εθνικέ πολιτικές ε, στήριξης αυτής της μετάβασης. Διότι διαφορετικά μπορεί να έχουμε ένα ε, ψηφιακό ε, χάσμα που θα σημαίνει ότι κάποιες αίθουσες θα κινδυνεύουν να καταργηθούν, να εξαφανιστούν. Αυτά είναι τα δύο ε, κύρια σημεία, ε, τα δύο σχέδια συμπερασμάτων, τα οποία θα υποβληθούν κατά το Συμβούλιο της 18ης Νοεμβρίου. Όσον αφορά την ε, εκπαίδευση και τα μίντια, ξέρετε ότι η γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου έχει μια μεγάλη παράδοση στην εκπαίδευση στα μίντια, που παίρνει πολύ συγκεκριμένες μορφές υπάρχει ε, θεσμοθετημένο ένα ανώτατο συμβούλιο για την ε, ε, εκπαίδευση στα μίντια και στις 2 και 3 Δεκεμβρίου θα οργανωθεί στο Βελικό Κοινοβούλιο ε, επ' ένα ε, συμπόσιο με θέμα εκπαίδευση για όλους. Θα συγκεντρωθούν εκεί όλοι αυτοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση στα μίντια στις Βρυξέλλες θα γίνει αυτό. Ε, σε αυτό το συμπόσιο ε, κάτι το οποίο θα τονιστεί είναι ότι η εκπαίδευση στα μίντια δεν θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στους νέους, που είναι φυσικά πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να αφορά και τους ενήλικες και όλους αυτούς που βρίσκονται εκτός του σχολείου. Πρόκειται για μια ε, μόνιμη, αν θέλετε, ή διαβίου εκπαίδευση στα μίντια. Αυτό είναι λοιπόν ένα συμπόσιο, συνέδριο που θα γίνει στις 2 και 3 Δεκεμβρίου τα κτίρια ε, εδώ του Κοινοβουλίου. Του Κοινοβουλίου, με συγχωρείτε, και όχι του Βελικού Κοινοβουλίου. Ε, και ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια επίσης, γιατί έγινε πολλής λόγο γι' αυτό, ε, για τις συμπαραγωγές. Οι συμπαραγωγές είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ περισσότερο για χώρες όπως το Βέλγιο που έχουν περιορισμένες δυνατότητες ε, παραγωγής. Χωρίς τις συμπαραγωγές δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κινηματογράφο, να κάνουμε κινηματογράφο. Αυτά ήταν τα ε, δύο-τρία λόγια που ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε ε, για τα πράγματα αυτά. ε, που μας ενημερώσετε για την παρουσία σας, γιατί δεν το ξέραμε στην αρχή της ακρόασης. Ε, <laughs> ζητώ συγγνώμη από την πολύ κυρία που είναι δίπλα σας, ε, που δεν της έδωσα το λόγο. Είμαι σίγουρη ότι θα δώσει τη μάχη της στο Συμβούλιο και στην Κορεπέρη για τις ιδέες που εξέφρασε ο συνάδελφός της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά που μας τα είπατε όλα αυτά έτσι όπως τα είπατε και άμα συνεχίσετε έτσι είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε έναν πολύ χρήσιμο ιτέρα σε εσάς. Για να τελειώσουμε, η κυρία Σίλβα από την Κομισιόν. Αβίβα Σίλβα, vous avez le Τα κατάφερα τελικά. Σας ευχαριστώ κυρία Πακ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την κυρία Πακ, διότι οργάνωσε αυτήν την σημαντική εκδήλωση. Και επίσης σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας ή στον κινηματογράφο που είναι ένα θέμα που με συναρπάζει πολύ και από ό,τι βλέπω και άλλους εδώ στο Κοινοβούλιο. Επίσης και όσον αφορά το βραβείο Lux και το πώς θα γίνει πιο δημοφιλές, πώς θα διαδοθεί στην Ευρώπη, όλα όσα κάνετε εκεί αποδεικνύουν τα λεγόμενα. Ήρθαμε εδώ από την υπηρεσία που ασχολείται με το media και θα γυρίσουμε στην βάση μας με πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και θα πρέπει να τα διερευνήσουμε ή στα πλαίσια του νέου προγράμματος Media, ε, αλλά και στα πλαίσια άλλων πολιτικών της ε, Κομισιόν. Είναι το θέμα το οποίο συνέχεια αναδύεται, δηλαδή το πώς θα αξιοποιηθούν τα διαρθωτικά ταμεία. Και αυτό το ακούσαμε σήμερα. Βεβαίως, ο κινηματογράφος είναι κάτι το μοναδικό. Δεν είναι μια κάποια βιομηχανία. Είναι κάτι που σχετίζεται ε, με την ταυτότητά μας, με εικόνες, με τα σενάρια, τις ιστορίες. Και θα πρέπει όμως να ξεχνούμε όμως το πόσος απασχολεί. Πόσοι εκεί βρίσκουν μια δουλειά και πόσο εκεί επίσης προκύπτουν ε, ε, ευκαιρίες εκμετάλλευσης της νέας τεχνολογίας. Γιατί αυτό το βλέπουμε για την είναι πάρα πολύ αληθινά. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ταυτόχρονα είναι μια σημαντική απειλή. Ότι δηλαδή η ψηφιακή επανάσταση είναι κάτι σαν 100 παλαιότερες επαναστάσεις, μια που καλύπτει το, το, το, το, όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις και αλλαγές από το, το βοβόγηματογράφο στην ομιλούντα, από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμα κλπ. και με κατανόηση του αναλφαβητισμού για τα μίντια και για το πρόγραμμα μίντια ασχολούμεθα και με χαρά άκουσα όλα όσα εξηγήσατε σήμερα. Πέντε χρόνια ασχολούμεθα με το θέμα το οποίο τώρα μόλις αρχίζει κάπως σε πολιτικό επίπεδο να συζητείτε είναι ένα εκ των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν για το νέο πρόγραμμα Media για να δούμε πώς θα συμπληρώσουμε το πρόγραμμα ό,τι του λείπει. Με δραστηριότητες, με εκδηλώσεις, με φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη. Και για να μην μακρηγορήσω, να σας πω ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε σε στενή συνεργασία στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Όποιος δεν έχει εμπλακεί, να ασχοληθεί. Και επίσης θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα, ούτως ώστε να πρεκοδοτείται όπως χρειάζεται ο κινηματογράφος για να ε, αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να διαδραματίσει το ρόλο που πρέπει. Και σας ευχαριστώ. Κύριε Σίλβα, σας ευχαριστούμε. Έχουμε τον πρόεδρο της Κομισιόν που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο του Βέντερς και των άλλων. Νομίζω και ελπίζω ότι έχει καταλάβει και μαζί με την κυρία Βασιλείου έχουν ευθυγραμμιστεί σε αυτή την πορεία. Αλλά θέλουμε και οι υπόλοιποι εκεί πέρα να καλύψουν αυτό που μας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα α, όλους εδώ, εδώ να τους ευχαριστήσω για τη συμβολή τους. Ε, ευχαριστώ όλους τους του συναδέλφου που συνεργάστηκαν. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και ευχαριστώ την Εκτελεστική Επιτροπή και να πω και δύο-τρία λόγια. Ο Βιβάνια είπε ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στην δύναμη της φαντασίας μας. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε η πολιτιστική ποικιλομορφία που έχουμε, που είναι μια πολυτέλεια, να γιορταστεί, να είμαστε ευτυχεί για αυτή. Να τη δώσουμε πνοή και ζωή, συζητώντας την, δείχνοντας ε, ταινίες σχετικές που θα τις δίνουμε και στα παιδιά. Και χαίρομαι που αναφέρθηκε το θέμα των σχολείων. Έχουμε το πρόγραμμα Κομένιους. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Κομένιους μπορεί πολύ καλά να ενταχθεί το θέμα αυτό. Στο νέο πρόγραμμα Κομένιους, αν μας ακολουθήσει η Εκτελεστική Επιτροπή, θα έχουμε το Κομένιους Teacher γιατί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα παιδιά εάν δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ε, διδάσκοντες πόσο σημαντική είναι μια ταινία ή ο κινηματογράφος γενικά. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το βραβείο Λουξ που, μας, που το αγαπάμε πάρα πολύ εδώ, μας δίνει τη δυνατότητα το βραβείο Λουξ να πάμε στα σχολεία. Εγώ με τους βραβευτές ε, ταινίες. Ε, φέτος μάθαμε με τις τρεις ταινίες που είναι οι τρεις από τις οποίες θα επιλεχθεί τελικά εκείνη που θα βραβευτεί, πηγαίνουν σε σχολεία, σε λύκεια και τους δίνουν κάποιες ιδέες τι σημαίνει παραδείγματο χάρη να ζει κανένας παράνομα, χωρίς ε, ταυτότητα ή τι σημαίνει μη, ένας φόνος τιμής πώς το ζει κανένας, πώς είναι αυτός της ε, ε, μια τουρκική οικογένεια. Γιατί αυτό είναι κάτι φρικτό που πραγματικά αγγίζει τη ζωή όλων και εκείνων που το ζουν απ' έξω και Και μετά μια γερμανοελληνική ε, ταινία που προσπαθεί να δείξει ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν την εντύπωση ότι απορρίπτουν τους υπόλοιπους στο μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και τελικά ανακαλύπτουν ότι και εκείνοι δεν είναι και διαφορετικά διαφορετικοί από τους άλλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Και όλοι οι συνάδελφοι, και εκείνοι που δεν είναι καν στην Επιτροπή Πολιτισμού, ότι με αυτούς τους, τις ταινίες μπορούμε πραγματικά να έρθουμε πολύ καλά σε επαφή με τα παιδιά και φέτος ε, η έδρα μας ας πούμε στην, ε, στην, ε, στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη, στο Μόναχο κλπ. δεν στέλνει απλώ κάποια φυλάδια έξω που το είπε ο Βιβέντες, σε μια κριτική σκληρή αλλά δίκαιη. <clears throat> Αλλά μπορούμε με τις ταινίες αυτές να πάμε στα σχολεία και να δείξουμε έτσι μια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τη γνωρίζουν και νομίζω ότι θα μονάχα με τη σήμανση των τροφίμων ε, σημαντικό και αυτό, αλλά το άλλο η επικοινωνία με την ταινία είναι πάρα πολύ σημαντική και γίνει τόσο πάει και πιο σημαντική. Και κάτι άλλο. Στο Κοινοβούλιο θέλουμε εμεί στι εξωτερικέ σχέσει, στη λεγόμενη υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην εξαφανιστεί ο, η πτυχή του πολιτισμού. Αλλά ακριβώ ε, μέσω αυτό να μπορέσουμε να προωθήσουμε ένα μήνυμα των ευρωπαϊκών μα πολιτισμών. Και αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μπορούμε να δράσουμε. Κατά τα άλλα θα φροντίσουμε το πρόγραμμα Media, το Media Μούντου στο καινούριο τώρα, να προωθηθεί όπως γίνεται τώρα, να έχει την ίδια πρικοδότηση, θα ήθελα να έχει περισσότερο, αλλά αυτό είναι θέμα του Συμβουλίου να μας διαθέσει τα χρήματα αυτά. Ε, μονάχα με κυριακάτικους λόγους και δεκάρικους δεν φροντίζουμε τίποτα για την Έντια δεν έκανε τίποτα ομιλίες και του λόγους, αλλά θα φροντίσει στην πράξη να έχει αποτελέσματα του χρόνου. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τις πολύ καλές ιδέες και λάψαρο που μας δώσατε. Μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι εμείς θα είμαστε ή θα παραμείνουμε ε, πρεσβευτές της ε, Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Ταινίας και μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Πέρα συνεδρίασής μας εδώ, η θα παραμεινουμε πρεσβευτες της ευρωπαικης κινηματογραφικης ταινιας και μπορειτε να βασιστειτε σε εμας περα συνεδριαση μας εδω η επομενη 17 Νοεμβρίου. forgot. I want to thank especially our Κοίταξε. Η... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία κύριε Βρυσόλη και τη Μαρή και τον Μπεατρό Πελιέ που εργάστηκαν πολύ σκληρά για το βραβείο Λουξ. Παρακαλώ σηκωθείτε να σας δούμε. Μαριφρό και η Μαρισέλα.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 Ευχαριστώ.